Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Κυρίες και κύριοι. Έχω τη χαρά ε, σήμερα να σας καλωσορίσω στο όνομα της Επιτροπής μας. Ε, πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν ε, να ασχοληθούμε πιο εντατικά με το σημερινό μας θέμα ε, θα παρακαλέσω τους προσκεκλημένους μας ε, να δείξουν κατανόηση που δεν είναι παρόντες πολλοί από τους ε, συναδέλφους ακόμα. Ελπίζω ότι θα έρθουν κατά τη διάρκεια της ακρόασης, αλλά καταλαβαίνετε έχουν και άλλες υποχρεώσει. Είναι ένα θέμα που ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, έχει γίνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η, ε, ο εφοδιασμός ενέργειας. Ε, και μάλιστα η, υπό διαφορετικές πτυχές ε, να έχουμε αρκετή ενέργεια, κατά πόσο θα είμαστε εξαρτημένοι από άλλες χώρες, πόσο μπορούμε να έχουμε ενέργεια ε, σε όσο γίνεται καλύτερες ε, τιμές για τους καταναλωτές μας, τους πολίτες μας και τέλος, εξίσου σημαντικό όμως πώς θα μπορούμε να έχουμε ε, ε, ενέργεια χωρίς ε, αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στο κλίμα. Είχαμε λοιπόν διάφορα νομοθετικά μέτρα. Όλοι Στην αρχή η συζήτηση εντό τη Ευρώπη, ήταν αρκετά εσωστρεφής. Ε, το θέμα ήταν η εσωτερική αγορά. Έχουμε προχωρήσει λίγο στο θέμα αυτό. Ε, πώς θα πετυχαίναμε ε, να έχουμε καλύτερες εντό εντός της Ευρώπης και αυτό είναι δύσκολο θέμα. Ο Επίτροπος Έτιγκερ προσπάθησε να ασχοληθεί με το θέμα. Μήπως όμως μέρος της λύσης είναι να κοιτάξουμε προς τα έξω, να δούμε μήπως υπάρχουν εκεί δυνατότητες, ευκαιρίες, ε, μήπως μπορούμε να βρούμε εκεί απαντήσεις ε, όχι μόνο σε θέματα ε, παροχής ενέργειας, ε, μήπως να κοιτάξουμε και τις γειτονικές μας χώρες και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Θέλουμε σήμερα να δούμε τι προγράμματα υπάρχουν στον χώρο της Μεσογείου, ποια είναι η κατάσταση, τι δυνατότητες ανάπτυξης υπάρχουν, πώς ε, ε, μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτό από πολιτικής, οικονομικής, τεχνικής πλευράς, ε, κοινωνικής πλευράς και... Ήδη αυτή τη βδομάδα είχαμε διάφορες ε, συζητήσει ε, για το θέμα αυτό. Ε, είδαμε ότι και τεχνολογικά δεν είναι πολύ απλό το θέμα. Προσπαθήσαμε όμως να διαφωτίσουμε τις διάφορες πτυχέ του θέματος και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέρφους που πήραν ε, την ε, πρωτοβουλία, που μας πίεσαν να κάνουμε αυτή την ε, εκδήλωση, αυτή την ακροασία. Αυτή ο ένας βρίσκεται, η μία βρίσκεται εδώ, η οποία έχει επιμείνει επανειλημμένα να έχουμε τη σημερινή ακρόαση, η Αγγέλικα Νίπλερ. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και τους εμπειρογνώμονες που έρχονται από κοντά και από μακριά, μάλιστα από πολύ μακριά έρχονται κάποιοι. Ελπίζω λοιπόν η σημερινή εκδήλωση να μας βοηθήσει και αυτούς που είναι εδώ σήμερα και αυτούς που θα μπορέσουν να διαβάσουν μετά τις ε, σχετικές πληροφορίες. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Ε, δίνω τώρα την Προεδρία στην Πρόεδρο του πρώτου πάνελ, την Αγγέλη Κανίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε Ρόιλ να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, και τους προσκεκλημένους μας. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να είμαστε εδώ σήμερα. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω, Χέρπερτ Ρόιλ, να ευχαριστήσω και τη γραμματεία που φρόντισαν για την πραγματοποίηση της σημερινής ακρόασης. Έχουμε πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Και στο πρώτο πάνελ έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές ε, που θα μας ε, παρουσιάσουν την, ηλική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, το πρόγραμμα Desertec. Ε, είναι και πάλι ιδιαίτερα επίκαιρο το θέμα αυτό, πόσο μάλλον που η Γερμανία σχεδιάζει την έξοδό της από την πυρηνική ενέργεια. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο γρήγορα τέτοια σχέδια. Ε, ε, θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τον Παουλ Φανσόν από την Τέσσερτεκ της Γερμανίας, τον κύριο Άλμπρετ Κάουπ από το med Είσαστε αλσα αυτός ε, στην ε, Βαρκελόνη ζείτε βέβαια ε, και να ευχαριστήσω τον Μάρκ Στρός που είναι ανώτατος σύμβουλος της Γραμματείας της Ένωσης της Μεσογείου. Και τέλος θα ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο Κρίστοφερ Μπούρχαρτ που είναι αντιπρόεδρος της First Solar. Χωρίς άλλα λόγια να δώσω τον λόγο στον πρώτο μας ομιλητή. Έχουμε προβλέψει το πολύ 10 λεπτά ανά ομιλητή για να ε, έχουμε χρόνο μετά και για την συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νίτλερ για την εισαγωγή αυτή. Κύριε Ρόιλ, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας ε, να μιλήσω εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή και πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιάσουμε το όραμα της ε, ΤΕΣΕΡΤΕΚ. Ε, να δούμε ποια θα είναι τα ε, επόμενα βήματά μας. Ο τίτλος είναι μια ε, σημαντική, ένα σημαντικό κίνητρο για την ε, μακροπρόθεσμη ευημερία της ε, Ευρώπης και θα σας παρουσιάσω τις διαφάνειες μου. Σίγουρα γνωρίζετε το την εικόνα της Ευρώπης και της Βορείου είναι λοιπόν η ιδέα της Desert Tech, οι περισσότεροι από εσά θα το έχετε ακούσει αυτό. Εκεί που υπάρχει πολύς ε, ήλιος και ε, λίγος κόσμος ε, στις ρήμους, εκεί που έχουμε η ηλιακή και ολική ενέργεια να την εκμεταλλευτούμε και για τον τοπικό πληθυσμό αλλά και για να μπορεί να γίνει μερικός τουλάχιστον εξαγωγή προς την Ευρώπη και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε αύριο μεθαύριο. Ε, αυτό θα διαρκέσει κάποιες δεκαετίες. Θα απαιτήσει λοιπόν ε, βαθμιαία ε, πρόοδο το θέμα αυτό. Ε, από τις ειδήσει θα γνωρίζετε ότι η Ευρώπη έχει μια περιφέρεια γειτονική, ε, την Βόρεια Αφρική. Τον τελευταίο χρόνο το <laughs> ανακαλύψαμε αυτό. Ε, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, πολύ φιλικοί και η Ευρώπη βλέπει εδώ χώρες ε, που βρίσκονται σε ε, φάση πολύ γρήγορης ανάπτυξης. Αυτό όμως απαιτεί και πολύ ενέργεια. Και σε κατά 85-90% η ενέργειά τους βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει γι' αυτό. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα ε, της Tech, δηλαδή εκεί που υπάρχουν οι πηγές ενέργειας ε, να τις εκμεταλλευτούμε. Η Ευρώπη ασχολείται με το θέμα της ενέργειας εδώ και αρκετό καιρό. Ε, προσπαθεί να πετύχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ε, στόχοι της είναι η αποτελεσματικότητα της ενέργειας, να μην υπάρχει σπατάλη, ε, πολύ καλή, ε, λογική χρήση της ενέργειας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το επόμενο βήμα είναι... να έχουμε αποκεντρωμένη ενέργεια. Κατόπιν υπάρχει η δυνατότητα στην ενέργεια ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών όταν κάποια ε, χώρα έχει περισσότερες πηγές εναλλακτικής ε, ενέργειας ε, να μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή. Και η Ευρώπη θέλει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπορεί να εισάγει και εναλλακτική ενέργεια από την ε, Μεσόγειο, από την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Ε, και οι τιμές αυτές θα είναι συμφέρουσες, ε, μάλιστα η τιμή θα είναι φθηνότερη από την μέση τιμή στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος εδώ. Η ευρωπαϊκή πολιτική, οι Βρυξέλλες έχουν κάνει πολλή δουλειά στο θέμα αυτό πριν ε, δύο χρόνια δημιουργήθηκαν κάποια ε, νομικά μέσα ε, η οδηγία για την ανταλλαγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά μας. Και επίσης να προβλέπεται η εισαγωγή εναλλακτικής ενέργειας από την Βόρεια Αφρική. Αυτό είναι το λεγόμενο άρθρο 9, ο ευέλικτος μηχανισμός και για την χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση των προγραμμάτων στη Βόρεια Αφρική. Αυτό θα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Και το μέσο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί, θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο ε, και ε, να μετατραπεί και σε πρακτικούς κανόνες και να υπάρχει κάποια εναρμόνιση ώστε όλοι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα αυτή. Πολύ βασικό στα προγράμματά μας ε, όσον αφορά την πραγμα... Ε, πραγματοποίηση ε, προγραμμάτων εναλλακτικής ενέργειας στην Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή Πολύ σημαντικό είναι όλα αυτά να γίνονται σε βάση εταιρικής σχέσης. Ε, πολύ σημαντικό παράδειγμα είναι το Μαρόκο. Ε, η συνεργασία μας με την μαροκινή κυβέρνηση και με την Μαζέν, την μαροκινή υπηρεσία ενέργειας, ε, βρίσκεται στο προσκήνιο. Αποτελεί πολύ καλή βάση όχι μόνο ε, για την ενέργεια αλλά και για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους. Δίδονται εδώ προοπτικές στον τοπικό πληθυσμό, θέσεις εργασίας, έχουμε μεταφορά τεχνογνωσίας κλπ. πολύ συγκεκριμένα. Ε, μεγάλο μέρος της ε, μακροπρόθεσμης ε, εργασίας μας ασχολείται με θέματα υποδομής. Ε, θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να ε, φροντίσουμε όλα αυτά να λειτουργούν και να δούμε ποιες είναι οι σημαντικές προκλήσεις. Μαζί με την ΜΑΖΕΝ έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα όπου στόχος είναι η παραγωγή 500 ΜΒ. Πρόκειται για, σχετικά, πρόκειται για πολύ μεγάλη εγκατάσταση ε, ε, ε, όταν μιλάμε για εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και θέλουμε να μειώσουμε και το κόστος της εγκατάστασης αυτής. Θέλουμε σιγά σιγά αυτή η εγκατάσταση που θα είναι πολύ ακριβή ε, σιγά σιγά να ενσωματωθεί στην αγορά και αποτελείται από δύο ε, μέρη. Ε, πρώτα θέλουμε μια εγκατάσταση με κάτωπτρα που προφανώς όλοι γνωρίζετε και μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. μιλάμε για 400 ΜΒ και 100 ΜΒ αντίστοιχα. δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. θα περάσω σε μια διαφάνεια που δείχνει πού ακριβώς βρισκόμαστε σε σχέση με την πολιτική και σε σχέση και με εσά. Ε, γνωρίζετε την ε, τεχνολογία αυτή και στην Ευρώπη, τα φωτοβολταϊκά, η βιομάζα, όλες αυτές οι τεχνολογίες ε, στην αρχή είναι πολύ ακριβές μέχρι να ενσωματωθούν στην αγορά. Εδώ αριστερά βλέπετε τις διαφορές ε, ανάμεσα στη δαπάνη και στην ε, αγορά. Στην αρχή είναι πολύ ακριβά τα προγράμματα αυτά, ε, χρειαζόμαστε λοιπόν στήριξη. Με τη στήριξη όμως και με στοχευμένες επενδύσεις στις χώρες της Βορείου Αφρικής που θα συμβάλλουν και με τη δική τους τεχνογνωσία Ελπίζουμε, ελπίζουμε οι εγκαταστάσεις αυτές να κινηθούν προς την κατεύθυνση της ε, αγοράς, να γίνουν δηλαδή οικονομικά συμφέροντα. Πιστεύουμε ότι αυτά τα προγράμματα κάποια στιγμή θα γίνουν ε, η βάση της ε, οικονομίας, η σπονδυλική της στήλη να το πούμε έτσι, διότι το κόστος μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ χαμηλό. Αυτή η μεγάλη πηγή θα ε, παρέχει μέρος ε, της ενέργειας. Τρία συγκεκριμένα βήματα προβλέπουμε και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο μας βήμα είναι επιτρέψτε μας να πραγματοποιήσουμε ε, το πρώτο πρόγραμμά μας. Ε, θα πρέπει η χρηματοδότηση ε, να διασφαλιστεί, να υπάρχει πολιτική υποστήριξη και να υπάρχει συνεργασία με τον σχετικό βιομηχανικό τομέα. θα πρέπει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Κατόπιν έχουμε το άρθρο 9, τον ευέλικτο μηχανισμό που σας ανέφερα. Θα πρέπει ε, να δοκιμάσουμε να δούμε εάν λειτουργεί. Ε, αυτό ως βοήθεια για τη χρηματοδότηση και όταν το πρώτο πρόγραμμα έχει δρομολογηθεί, τότε στα πλαίσια μιας ε, μακροπρόθεσμης ε, εταιρική σχέσης ανάμεσα στην Ευρώπη και την ε, Βόρεια Αφρική, να βρούμε ποια στοιχεία είναι σημαντικά για την Ευρώπη και για τη Βόρεια Αφρική. η ενέργεια, για παράδειγμα, πιθανότατα και άλλα πράγματα, αλλά εγώ αναφέρομαι κυρίως στην ενέργεια. όχι μόνο στο Μαρόκο, αλλά και στην την Ισία, στην Αίγυπτο, σε άλλα μέρη ενδεχομένως ε, εξετάσουμε τα θέματα αυτά της ε, ενέργειας. Ε, ελπίζουμε ότι αυτά θα οδηγήσουν σε, θέση, σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης κλπ. Ε, τέλος, κλείνοντας να πω ότι ήθελα να σας προσκαλέσω σε μια διάσκεψη που οργανώνουμε φέτος στο Κάιρο, όπου θα είναι παρόντες πολύ πολύ ε, πολιτικής επίπεδο λήψη αποφάσεων και ο κύριος Έτιγκερ είπε ότι θα συμμετάσχει. Ε, θα συμμετάσχουν ε, άνθρωποι από την Ευρώπη και από την Βόρεια Αφρική, Υπουργοί και άλλοι. Σας προσκαλούμε θερμά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίασή σας και για την πρόσκληση στη διάσκεψη στο Κάιρο. Αυτό σίγουρα θα, το, ε, ε, θα εξετάσει ο πρόεδρος μαζί με τους ε, συντονιστές την δυνατότητα συμμετοχής μας με ειδική αποστολή. Χωρίς πολλά πολλά θα παρακαλούσα τον επόμενο μιλητή, τον κύριο Κάουπ, να ξεκινήσει την παρουσίασή του. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Λέγομαι Άλμπρεχτ Κάουπ, και τρία χρόνια μένω στο Κάιρο της Αιγύπτου. Συντονίζω και ε, ε, ρυθμίζω τον διάλογο με τις νότιες γειτονικές χώρες όσον αφορά ε, την, ε, την ηλεκτρική ενέργεια. Θα ήθελα σήμερα δηλαδή ε, να σας μεταφέρω αυτό που ήδη μας λένε εμάς εδώ και τρία χρόνια σχετικά με τις ευρωπαϊκές μας ιδέες. Ε, να ε, ενσωματωθεί δηλαδή η αγορά ενέργειας της Βορείου Αφρικής στην Ευρωπαϊκή. στο εγγύς μέλλον να υπάρχει εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι καθήκον μας ε, στα πλαίσια ενός ε, προγράμματος της ε, Κομισιόν. Θέλουμε να είμαστε καταλήτης. σε πέντε τόμους που εκδόθηκαν πριν ένα εξάμεινο περίπου, που μπορείτε να βρείτε και στο, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια. Ε, σε αυτούς τους πέντε τόμους λοιπόν παρουσιάζουμε ε, τον ε, ενεργειακό τομέα στην Μεσόγειο. Τι λύσεις υπάρχουν, πώς μπορεί να κλείσει ε, ο περίφημος δακτύλιος, πού υπάρχουν ε, δυνατότητες, τι οικονομικές δυσκολίες υπάρχουν. Και τι ε, νομικά και διοικητικά εμπόδια υπάρχουν στην εξαγωγή της ηλιακής ενέργειας. Για καθέναν από αυτούς τους πέντε τόμους θα σας πω απλά λίγα λόγια. Ε, πραγματικότητα ε, σε σχέση με τα οράματα. Δύο ε, Δύο πτυχές υπάρχουν εδώ. Αριστερά βλέπετε ένα μεγάλο ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι πολύ σαφές τι μπορεί να γίνει Σήμερα με την υπάρχουσα τεχνολογία ε, βλέπετε όμως ότι ήδη στη Λιβύη σταματάει το ναι. Ε, συμπεριλαμβάνονται εδώ το Μαρόκο, η Αλληλεργία, η Ισία. Βλέπετε και δύο νούμερα, 5% και 9% τα οποία σας δείχνουν ότι ε, η περιφέρεια αυτή παίρνει ενέργεια από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει αρκετή ενέργεια εδώ. Αυτό ήθελα να το τονίσω. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση. Στα δεξιά της κίτρινης γραμμής, εκεί που ξεκινάει η Αιγυπτός, κατά τη γνώμη μου, δεν θα υπάρξει άμεση σύνδεση μέσω της Μεσογείου θα μπορούσε να φτάσει κανείς στην Κρήτη ή στην Ελλάδα. Ε, αλλά θα λέγαμε ότι με τις ε, υπάρχουσες τεχνολογίες ε, μπορούμε να πούμε ναι στην αριστερή πλευρά του χάρτη, όχι όμως στη δεξιά. Είναι πολύ μεγάλα τα περάσματα. Βλέπετε και τις δύο παχές μαύρες γραμμές. Ο κύκλος σχεδόν έχει κλείσει βλέπετε ότι στην, ε, στα Συριακά σύνορα έχουμε φτάσει μέχρι εκεί έχουμε φτάσει θα σας το εξηγήσει αυτό ο Μάνιουελ και βλέπετε τις ε, δύο μαύρες γραμμές κάτω στη Λιβύη, στη Λιβύη ε, εδώ και 10 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε. Από το Μαρόκο λοιπόν δεν μπορούμε να στείλουμε ενέργεια προς τη Συρία, Συρία. Δεν έχουν γίνει δύο προσπάθειες ε, τα τελευταία δέκα χρόνια, έχουν αποτύχει όμως. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα όσον αφορά την εξαγωγή και την ε, ανταλλαγή ε, ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο. Αν Σκεφτείτε ποιες είναι οι ανταγωνιστικές ε, πηγές ενέργειας ε, στην ηλιακή ενέργεια ε, και στη φωτοβολταϊκή. Ο ανταγωνιστής μας είναι το φυσικό αέριο. Δεν είναι ούτε τα ορυκτά καύσιμα, ούτε κανένα άλλο. Αριστερά ε, βλέπετε, ήθελα να σας δείξω το, κάος, ε, το χάος στην ε, τιμή του αερίου. Βλέπετε τι διακυμάνσεις έχει η τιμή του φυσικού αερίου. Ανάμεσα σε 5 και 15 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του εδώ και πολύ καιρό. Εάν συλλέξετε στοιχεία από τους συνομιλητές μας στις ε, εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος. Ε, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα δούμε διπλασιασμό, θα δούμε διπλή ε, κατανάλωση αερίου, πετρελαίου και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Εμείς όμως είχαμε ελπίσει να τετραπλασιάσουμε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. και η υδροελεκτική ενέργεια θα μειωθεί ε, στο μισό ε, ε, ως προς το ποσοστό διότι δεν υπάρχουν νέες εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο. Θα πρέπει λοιπόν να αντισταθμίσουμε την κατάσταση αυτή. το μεγαλύτερο εμπόδιο, όμως, ε, εμπόδιο μας ε, και θα ήθελα να το αναφέρω αυτό. Είναι το γεγονός ότι ε, αυξάνεται ραγδαία η, ζήτηση ρεύματος κατά 10-11% το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παράγουμε μόνοι μας ε, την ε, απαραίτητη ενέργεια, εξαρτιόμαστε από την Ευρώπη. Και κάθε συνομιλητής μας λέει γιατί να αγοράσω ηλιακή ενέργεια αφού στοιχίζει 5 με 10 φορές περισσότερο κεφάλαιο, όχι κόστος παραγωγής. Μας λένε ότι έχουμε άλλα προβλήματα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε αρκετή ενέργεια. Και υπάρχει εδώ και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους ε, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ενέργειας ε, θα πρέπει να είναι κατά 5 με 10% πιο ακριβό το ρεύμα τους ε, για να ε, καλύψουν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Είναι λοιπόν πιο ακριβή η ιδιωτική παραγωγή ενέργειας. Θα ήθελα να σας δείξω εδώ την διαμόρφωση των τιμών που θα είναι σημαντική για μας. Έχουμε χωρίσει ε, στα δύο τις ε, χώρες. Βλέπετε τις κίτρινες με την Αίγυπτο. Ε, εδώ έχουμε 3,8 με 2,5 Η κίτρινη ομάδα βρίσκεται στα 7 cents. Το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Τινησία και βλέπετε ε, στο ΜΟΦ κουτάκι ότι η αιωλική ενέργεια είναι ε, πολύ ε, συμφέρουσα εδώ. Οι κίτρινες χώρες είναι συγκρίσιμες με τις τιμές στην Ευρώπη. ενώ βλέπετε το, το πάνω μέρος, το 23 με 38 cents, είναι οι τιμές του οικιακού ρεύματο στην Ευρώπη. Το 23 με 38 cents και κάτω 14 με 23 ε, cents ε, είναι οι τιμές παραγωγής ε, του, του ηλιακού ρεύματο, Σε παρένθεση βλέπετε πόσο θα στήχιζε σε έναν ε, ιδιώτη παραγωγό ενέργειας, σε ιδιωτική επιχείρηση παραγωγής ενέργειας ε, τις τιμές. Ε, οι τιμέ εδώ πρέπει να είναι υψηλότερε για να καλύψει ενδεχόμενου κινδύνους. Αυτό σημαίνει ότι ανταγωνιστική είναι μόνο η αιωλική ενέργεια και τέσσερις χώρε έχουν αρκετά χαμηλέ τιμές ώστε να πρέπει να επενδύσουμε πολλά χρήματα για να γίνει ανταγωνιστική. Και τώρα οι καλές ειδήσει. Παρόλα αυτά, εάν σήμερα θέλατε να δημιουργήσετε μια εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας σε 500 ΜΒ και θα θέλατε σε 20 χρόνια να δείτε αν έχετε λάβει τη σωστή απόφαση, θα πρέπει να Πείτε ναι, διότι βλέπετε εδώ ε, το, ε, τα πράσινα νούμερα, είναι το κέρδος. Ε, στην αρχή βλέπετε πόσα πρέπει να πληρώσετε στην αρχή. Το, οι πράσινες γραμμές είναι το κέρδος. είναι λοιπόν συγκρίσιμη η κατάσταση με, είναι σε σύγκριση με τις αυξανόμενες τιμές ε, του αερίου και, ε, και του πετρελαίου. Βλέπουμε ότι συμφέρει πιο πολύ ε, αυτού του είδους η επένδυση, παρότι στην αρχή έχουμε ε, αυτές τις κόκκινες γραμμές. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι αυτό που βλέπετε αριστερά, όπου οι κόκκινες γραμμές δεν ε, μικραίνουν καθόλου. Ε, να μην διαλέξουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο. Εάν έχουμε μια εγκατάσταση όπου μετά από 7 με 10 χρόνια ε, υπάρχει κέρδος και ε, από την οποία υποφιλείται όλη η κοινωνία, αυτές είναι οι χρήσιμες εγκαταστάσεις. Και φτάνω τώρα στο καυτό θέμα των εξαγωγών. Πριν δύο χρόνια Ακούσαμε δηλώσεις από την Ευρώπη ότι η Ευρώπη χρειάζεται την ηλιακή ενέργεια. Αυτό δεν μας βοήθησε πολύ διότι ο καθένας εδώ και τρία χρόνια μας λέει ότι «Ε, χρειάζεστε το ηλιακό, την ηλιακή μας ενέργεια αλλά τίποτα δεν γίνεται. Εάν ε, Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Βλέπετε εδώ ε, τις ε, δικές μας τιμές, το hour tariff, 26 ε, cents, 26 λεπτά. Εάν χτίζαμε εγκαταστάσεις στο νότο, έχουμε σαν να λέμε δύο ήλιους σε σχέση με από πάνω. Έχουμε την διπλάσια ηλιακή ενέργεια, ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να ε, έχουμε τιμή 20 λεπτά. Ε, συγγνώμη, 13 ε, cents. Ε, δεν μπορούμε να χτίσουμε πιο φτηνά τις εγκαταστάσεις. Υπάρχει όμως περισσότερος ήλιος και ναι, θα πρέπει να μεταφέρουμε την ενέργεια μετά για την εξαγωγή. Αυτό μπορεί να στοιχήσει το 10%. Αυτό σημαίνει ότι επί της αρχής η τελική τιμή θα είναι 20,3 ε, λεπτά. Οικονομικά λοιπόν αυτό θα ήταν πολύ λογικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν ε, επενδυτές στο Νότο, διότι δεν υπάρχουν αγοραστές στο Βορρά. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Ε, εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας χτίζει κανείς μόνο αν, έχει, αν ξέρει ότι έχει κάποιον πελάτη για τα επόμενα 20 χρόνια. Τρεις ε, τεχνολογίες ουσιαστικά είναι ανταγωνιστικές. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις ότι ε, οι ε, μονάδες παραγωγής με αποθήκευση συσσωρευμένη ηλιακή ενέργεια δηλαδή ότι είναι αξιόπιστες, δεν έχουμε πρόβλημα ε, ούτε με την αιωλική ενέργεια και ε, βλέπουμε ότι και οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ουσιαστικά έχουν κερδίσει ε, σε σχέση με την συσσωρευμένη ηλιακή ενέργεια λόγω του κόστους. Αυτό σημαίνει ότι η φωτοβολταϊκή τεχνολογία πολύ γρήγορα θα φτάσει και την αιωλική ενέργεια. Σε τρία-πέντε ε, χρόνια μπορεί να γίνει και ανταγωνιστική σε σχέση με την ε, αιωλική ενέργεια. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Πέντε συστάσεις έχουμε. με βάση του, το, το υψηλό επενδυτικό κόστος, όχι το κόστος παραγωγής, είναι σημαντικό ε, να ε, συμμετάσχουν μεγαλύτερα ταμεία και τράπεζες. Οι αραβικές τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν ε, πολύ συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση, τη ζήτηση, τη ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική ε, η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, ιδιαίτερα για τις ε, πηγές. Επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο βορρά, να βρούμε αγοραστές ε, που να, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε το άρθρο 9 και θα πρέπει να ε, καταλήξουμε σε ένα μείγμα πρασίνων και ορυκτών πηγών ενέργειας, διότι αλλιώς ε, δεν ε, θα συμφέρει οικονομικά ε, η όλη κατάσταση. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά την ικανότητα, το δυναμικό των εγκαταστάσεων αυτών. Θα πρέπει δηλαδή να εξετάσουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης και η τελευταία μου διαφάνεια ε, είναι αυτή που βλέπετε. Εγώ, Εγώ μένω στην ε, Αίγυπτο. Εάν εάν θέλαμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με ε, με ανθρώπους ε, θα στήχιζε από 25 μέχρι 2,5 ευρώ ανά κιλοβατόρα όπως βλέπετε αν έτρεχε ο κόσμος ανάλογα βέβαια και με το τι τρώνε αν τρώνε ε, χαμπουργκερ ή ε, ελαιόλαδο. Ε, πάντως ούτως ή άλλως σε συμφέρουν οι, ανα, εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Νίπλερ. Θα δώσω το λόγο στον τελευταίο μας ομιλητή τον κύριο Στράου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και μένα στην συνάντηση αυτή και έτσι έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω το τι γίνεται από πλευρά της Ένωση για την Μεσόγειο, της Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο στον τομέα της ενέργειας και τη ηλιακή ενέργεια. Έχουμε το Μεσογειακό Ηλιακό Σχέδιο για την Μεσόγειο είναι μία από τις έξι προτεραιότητες που έθεσαν οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων στη διάσκεψη των Παρισίων τον Ιούλιο του 2008. Στη συνέχεια, μπήκαμε περισσότερο σε λεπτομέρειες. Καθορίσαμε στόχους που είναι η ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο της ηλιακής δηλαδή, παρά την ονομασία του σχεδίου που είναι Mediterranean Solar Plan. Μιλήσαμε λοιπόν για 20 επιπλέον γίγαβατ. Παραγωγή. Ε, δεν μιλάμε για την εξαγωγή, μιλάμε για την παραγωγή. Γιατί η εξαγωγή είναι ένα τμήμα το οποίο θα καθοριστεί αργότερα. Είχαμε σκεφτεί ότι ίσως είναι το 1 τέταρτο των 20 αυτών ε, γιγαβάτ. Για να πετύχουμε όμως αυτό το στόχο, οι χώρες ε, μέλη θελήσαν να εκπονηθεί ένα master plan προκειμένου να διευκρινιστούν ακριβώς τα μέσα με τα οποία θα πετυχαίναμε το στόχο μας. Πρόκειται λοιπόν για μια μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία ευρωμεσογειακή, η οποία εγγράφεται στα πλαίσια τα γενικότερα παγκόσμια και ευρωπαϊκά στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που γίνονται για την καταπολέμηση της αλλαγή του κλίματος και στα πλαίσια των ε, πρωτοβουλειών που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα του 2020 Και πέρα από την δήλωση των Παρισίων έχουμε και την δημιουργία της γραμματείας, η οποία στην ουσία υπάρχει από πέρυσι μόνο. Στο μεταξύ όμως έχουν συμβεί πολλά. Έχουμε εθνικές στρατηγικές οι οποίες εγκρίθηκαν σε πολλές μεσογειακές χώρες, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τινησία αλλά και σε άλλες χώρες. Έχουμε επίσης βιομηχανικές πρωτοβουλίες, Belgrid, Τεσσευτέ κλπ. Και έχουμε επίσης και νέα οικονομικά μέσα από τα διάφορα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι λοιπόν τα τελευταία αυτά δύο χρόνια έχει προχωρήσει μια διαδικασία, καταλητική θα έλεγα, που ξεκίνησε από τη δήλωση των Παρισίων, που έδωσε νέα όθηση σε όλα αυτά. Στα πλαίσια λοιπόν της δήλωσης των Παρισίων, η Γραμματεία της Ένωσης για την Μεσόγειο ανέλαβε την ευθύνη απευθείας και φαίνεται αυτό στο παράρτημα της δήλωσης των Παρισίων να ασχοληθεί με τη σκοπιμότητα της δημιουργίας και της εκμετάλλευσης ενός ε, τέτοιου σχεδίου ηλιακής ενέργειας για την Μεσόγειο. Η εντολή αυτή επιβεβαιώθηκε και από τους εκπροσώπους των 43 χωρών που ζήτησαν από την γραμματεία μας να συντονίσει τη δημιουργία αυτού του master plan σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και το σύνολο των συμμετοχόντων και των ενδιαφερομένων. Για το σκοπό αυτό η γραμματεία θα βασιστεί πρώτα απ' όλα στο κεκτημένο που έχουμε τα δύο τελευταία χρόνια και στα έγγραφα στρατηγικής σημασίας που έχουν υιοθετήσει προηγουμένως τα κράτη-μέλη, πριν δηλαδή από τη δημιουργία της γραμματείας μας. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση στις Βρυξέλλες με όλους τους ενδιαφερόμενους εδώ και μερικούς μήνες, το Φεβρουάριο έγινε αυτό. Τι θα προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε βάσει αυτών είναι δύο-τρία πράγματα τα οποία είναι τα μεταξύ τους και τα οποία είναι ζωτική σημασία και είναι ζωτική σημασία να τεθούν σε εφαρμογή συγχρόνω. Το ένα είναι ο στόχο του master plan, που είναι όσο γίνεται με μεγαλύτερη συνένεση να φτιάξουμε ένα πλαίσιο αναφορά με όλου του ενδιαφερόμενου και κυρίω με τα κράτη-μέλη. Αυτό το πλαίσιο αναφορά θα μα επιτρέψει μαζί να βρούμε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε βασικά στοιχεία κλειδί. Μερικά από αυτά ανέφεραν ήδη οι προλαλήσαντες. Τα στοιχεία αυτά είναι βασικά γιατί από αυτά εξαρτάται η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας και αναλλακτικών πηγών ενέργειας στην Μεσόγειο αλλά και όχι μόνο. Πρέπει λοιπόν μαζί να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ποια είναι τα νομοθετικά πλαίσια, τα αριθμιστικά, τα μέσα χρηματοδότησης, υποδομές, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί, η μεταφορά ε, know-how επίσης, η ανάπτυξη ικανοτήτων. Όλα αυτά είναι κεντρική σημασία ε, και αποτελούν μέρος του ε, Μεσογειακού Solar Plan και θα χρησιμοποιήσουν μελέτες που έχουν ήδη γίνει, δεν χρειάζονται νέες. Έτσι, στα τέλη του 2012 πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε θέση να θέσουμε ένα έγγραφο πως ε, έγκριση στη, στους υπουργούς. Εννοείται ότι δεν πρέπει να περιμένουμε το 2012 και 2013. Στο μεταξύ πρέπει να εντοπίσουμε και να στηρίξουμε συγκεκριμένα πιλωτικά προγράμματα αναπτύσσοντας νέα οικονομικά μέσα για να προχωρήσουν τα σχέδια και τα προγράμματα αυτά. Αυτά είναι τα καθήκοντα λοιπόν που αναλαμβάνουμε και που ελπίζουμε να φέρουμε και σε πέρας. Ποια είναι η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε. Η γραμματεία αποτελεί βασικά μια πλατφόρμα και έχει περιορισμένα μέσα στη διαθεσή της. Ο ρόλος της είναι να αποτελέσει ένα σημείο όπου συναντιόνται διάφορες ιδέες και δράσεις. Έπειτα πρέπει να υπάρχει πολιτικός έλεγχος για τα θέματα που χειριζόμαστε είναι ευαίσθητα πολιτικά. Άρα θέλουμε, όπως έλεγα και πριν, να έχουμε μία κοινή άποψη, να συγκεντρώνουμε δηλαδή μία κοινή θέση μεταξύ διαφόρων χωρών μελών. Δηλαδή εμείς είμαστε ουδέτεροι. Οι χώρες εκατέρωθαν της Μεσογείου ε, μαζί θα αποφασίσουν. Εμεί από μόνοι μα είμαστε ουδέτεροι και δεν έχουμε κανένα συμφέρον υπέρ τη μια ή της άλλης τεχνολογίας. Εννοείται λοιπόν ότι θέλουμε τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, των πρώτων μελών δηλαδή καταρχήν, τη βιομηχανία, των θεσμικών οργάνων αλλά και τη κοινωνία των πολιτών. Με το master plan αυτό θέλουμε, αλλά εδώ βέβαια θα το συζητήσουμε ξανά με τα κράτη-μέλη, θέλουμε να προχωρήσουμε στα πέντε κύρια σημεία τα οποία αναφέρθηκαν και πριν. Πρώτον, πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεύτερον, χρηματοδότηση. Τρίτον, υποδομές, φυσικές υποδομές. Τέταρτον, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν ως καταλύτες στη βιομηχανία. Και τέλος, μεταφορά know-how και ε, οικοδόμηση ικανοτήτων. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τους εταίρους μας, να δούμε ποια είναι η δομή αυτών των ε, στοιχείων. Το πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο τι είναι. Είναι δέσμευση πολιτική που αναλαμβάνουν οι χώρες μέλη για να προσφέρουν ένα πλαίσιο αναφοράς που θα επιτρέψει στους επενδυτές να ξέρουν που πάνε. Αλλά πρόκειται για την ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα ευνοεί την ανάπτυξη των ανασώσιμων πηγών ενέργειας. Και έτσι πάλι θα αποτελέσουν καταλήτη για επενδύσεις ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο οι ανανώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλήσαμε και για τη χρηματοδότηση. Οι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν στο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη χρηματοδότηση για ηλεκτρισμό, στις ανώσιμες πηγές και στα ε, ορυκτά. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε καλύτερες λύσεις. Τα μέσα Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα. Αναφερθήκαμε στο άρθρο 9. Αποτελεί ένα σημαντικό μέσο, πράγματι. Όμως πρέπει να υπάρχει ισορροπημένη παραγωγή, τόσο για την τοπική ε, χρήση, όσο και για τις εξαγωγές. Δεν έχει νόημα να γίνονται μεγάλες εξαγωγές, γιατί χρειάζονται ηλεκτρισμό και οι ίδιες οι χώρες νοτίως της Μεσογείου. Το άρθρο 9, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, έχει οδηγήσει στο να χυθεί πολύ μελάνι. Τώρα χρειαζόμαστε μια πολιτική δέσμευση από τους μελλοντικού ε, Ευρωπαίους, ευρωπαϊκούς μάλλον πελάτες, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ένα άλλο μέσο που ήδη υπάρχει και που έχει να κάνει με την οικονομία του άνθρακα, είναι ένα στοιχείο ανησυχία για τη σημερινή κατάσταση μπορεί να μας οδηγήσει στο να πάμε πίσω αντί να προχωρήσουμε. Ακόμα και αν καλύπτει ένα περιορισμένο κομμάτι, ένα μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους του σχεδίου για τις αναλλακτικέ ε, ενέργειες, δυστυχώς υπάρχει μια διάταξη της ε, οδηγίας ΙΤΕΣ που λέει ότι για προγράμματα τα οποία πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2012 δεν αποτελούσαν ε, σημείο αναφοράς, η πιστοποίηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο αν υπάρχει διμερή συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την χώρα αμφιτριώνα. Προ το παρόν δεν υπάρχει καμία όμω τέτοια χώρα, τίποτα δεν έχει γίνει. Πράγμα που σημαίνει ότι παρόλο που προσπαθούμε να αναπτύξουμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών της Μεσαιγείου, κινδυνεύουμε σε λίγου μήνε να έχουμε χάσει 4 με 5% του PSM, γιατί αν δεν έχει γίνει τίποτα δεν θα έχουμε πιστώσει για τον άνθρακα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα αυτά. Κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε επίσης να μειώσουμε και τον κίνδυνο. Γιατί αναφέραμε τις ανώσιμες πηγές ενέργειας φυσικά, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με μηχανισμούς οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε το κόστος. Σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι χρηματοδότηση υπάρχει. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα, τα οποία να τα συντονίσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί. μονομένα, κανένα οικονομικό μέσο ή άλλο μέσο δεν μας βοηθάει να λύσουμε το πρόβλημα είναι ένα σύνολο μέσων που πρέπει να διαρθρώσουμε μεταξύ του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Χρειάζεται πολιτική απόφαση, χρειάζεται πολλή δουλειά και πολλή συνεργασία. Αν δεν τα καταφέρουμε, δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε σε μεγάλη κλίμακα την ε, τεχνολογία αυτή που θέλουμε. Και όπως υπενθύμησε και ο συνάδελφο, αν δεν αναπτυχθεί η τεχνολογία αυτή σε μεγάλη κλίμακα, δεν θα πέσει το κόστο, άρα δεν θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Ένα θέμα είναι τα δίκτυα υποδομών. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί αυτά θα τα ακούσουμε και από άλλες παρουσιάσεις. Πρέπει όμως να έχουμε μια σφαιρική εικόνα των υποδομών και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο θέμα της διασύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών της Μεσογείου, που είναι κεντρικό θέμα, αλλά πρέπει να δούμε και τις διασυνδέσεις νοτίως της Μεσογείου, όπως υπενθύμησε ο συνάδελφος. Και πρέπει να δούμε και την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ χωρών που βρίσκονται νότια της Μεσογείου, ώστε ο πράσινος ηλεκτρισμός να φτάσει και στην Ευρώπη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αποτελέσουν ε, ε άνισμα ανάπτυξης για τις χώρες νοτίως της Μεσογείου. Δεν θέλουμε μαζικές εισαγωγές από τις βόρειες χώρες. Όχι, θέλουμε να αναπτυχθούν οι χώρες νοτίως της Μεσογείου και να βρούμε τρόπους γι' αυτό. Μήπως πρέπει να έχουμε ρήτρε που να αναφέρονται σε αυτό, όπως συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις, να προβλέψουμε μέτρα ειδική στήριξης, να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες έρευνας με χρηματοδότηση από την πλευρά μας. Όλα αυτά είναι ιδέες. Το βέβαιο είναι ότι 30 με 50% είναι η συμμετοχή των ε, χωρών ε, θεωρητικά, αλλά δεν πάνε πάνω από 20%. Οπότε κινδυνεύουμε να ταράξουμε το ισοζύγιο στις χώρες αυτές. Πρέπει επίσης να δουλέψουμε πολύ και στο θέμα της μεταφοράς know-how και οικοδόμησης ικανοτήτων. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό. Υπάρχουν πολλοί που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να βρεθούν οι σωστές πλατφόρμες για να γίνει αυτό. Να λοιπόν θέματα που πρέπει να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη για να μπορούμε να είμαστε ρεαλιστές και για να καταλήξουμε σε μια συνενετική πρόταση. Η δουλειά είναι τεράστια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να πιέσουν και να δουλέψουν καταλητικά. Για να ολοκληρώσω, Θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Τα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα είναι ζωτική σημασία. Θα τα καταφέρουμε, ελπίζω. Γιατί έχουμε πολλά ατού για να το πετύχουμε. Υπάρχει και πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Υπάρχει επίσης και το θέμα της ε, ασφάλειας εφοδιασμού όσον αφορά την ενέργεια. Άρα έχουμε κάθε συμφέρον να προχωρήσουμε από κοινού όλες ε, οι χώρες ώστε και οι μεσογειακές χώρες να μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι εξελίξεις τρέχουν, είτε πρόκειται στην Νότια Αφρική, είτε πρόκειται για την Ινδία, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε αυτό. Και αν τα πράγματα δεν γίνουν στις χώρες της Μεσογείου που έχουν τόσο μεγάλα ατού, τότε άλλες χώρες θα πρωταγωνιστήσουν και δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα του αυτά που έχουν και το συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ε, ευχαριστώ θερμά και για την ε, δική σας ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Να δώσω τον ε, λόγο στον κύριο Μπούρκχαρτ να ξεκινήσει και εκείνο ε, την ομιλία του. Ευχαριστώ πολύ. Ενώ περιμένω να εμφανιστούν οι διαφάνειες. Ανάμαστε. Μία σύντομη εισαγωγή για όσους από εσά ε, δεν γνωρίζετε την First Solar. Είμαστε μία εταιρεία ηλικίας 12 ετών, σχετικά νέα δηλαδή, αλλά σχετικά ηλικιωμένη στον ε, τομέα αυτών. Έχουμε έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε όμως ε, μεγάλη ε, παραγωγική μονάδα στις, στη Γερμανία, τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Μαλαισία, ενώ σχεδιάζουμε μονάδες παραγωγής στην Γαλλία και το Βιετνάμ. Είμαστε ε, δεύτερη εταιρεία παραγωγής στον κόσμο ε, στα φωτοβολταϊκά και η μεγαλύτερη ε, στις μονάδες λεπτής μεμβράνης. Και έχουμε το χαμηλότερο κόστος για τα φωτοβολταϊκά αυτή τη στιγμή, 75 cents του δολαρίου αναβάτ αυτή τη στιγμή. Ε, δεν θα πω σε πολλές ε, λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να σας πω ε, για τις μονάδες που έχουμε φτιάξει σε ρυθμικέ περιοχές. Έχουμε την μεγαλύτερη τέτοια εγκατάσταση στον κόσμο, 2,4 γιγαβάιτ μέγεθος. κοιτώντας ε, την ε, περιοχή ΜΕΝΤΑ, της Μεσογείου δηλαδή, ε, Πιστεύω ότι τα φωτοβολταϊκά αποτελούν μεγάλη ευκαιρία και αν θέλει να οικοδομήσει κανεί γρήγορα δυναμικό τα φωτοβολταϊκά και γενικά η ηλιακή ενέργεια αποτελεί σημαντική ευκαιρία. Προφανώς υπάρχει και η δυνατότητα για πιο αποτελεσματική διαχείριση των όσων υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή. Συνεργαζόμαστε με ε, ανθρώπους που ήδη ε, κινούνται στον τομέα της ενέργειας για να αναπτύξουν ε, έναν φάκελο με μεγάλο ποσοστό ηλιακής ενέργειας. Γενικά υπάρχει ανάγκη για αύξηση της ε, παραγωγής ε, ηλεκτρικής ενέργειας ε, στη Μεσόγειο και νομίζω ότι είναι ένας από τους τομείς όπου ειδικά τα φωτοβολταϊκά που μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά στην ζήτηση είτε με τρόπο συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο προσφέρει πολλές δυνατότητες. Επίσης όταν μιλάμε για την ε, η οικοδόμηση υποδομής για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα πρέπει να γίνει ε, σε τοπικό επίπεδο. Μπορούμε να αποφύγουμε τις ε, απώλειες λόγω της μεταφοράς και της κατανομής εάν χτιστούν έξυπνα οι μονάδες. Επίσης, όσον αφορά την δημιουργία θέσεων εργασίας, μία μία ε, μονάδα, ε, μία ομάδα ε, εργατών χρησιμοποιεί 275 εργαζόμενους την ημέρα, εργάτες την ημέρα για κάθε μεγαβάτ. μιλάμε δηλαδή για πολλές θέσεις εργασίες. Επίσης σημαντικό είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας. σίγουρα πολλά έχει μάθει ο τομέας και η μεταφορά της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων είναι κάτι πολύ σημαντικό στον τομέα αυτόν. Μας ενδιαφέρουν επίσης όχι μόνο οι περιβαλλοντικές πτυχές, ε, οι ενεργειακές πτυχές, αλλά και οι περιβαλλοντικές. Ε, επίσης, ε, σημαντικό στοιχείο είναι και οι σημαντικές δεκιμάνσεις στι τιμέ. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι εικόνα έχουν αυτές οι μεγάλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και ούτε ξέρουν τα πλεονεκτήματά τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν χρησιμοποιούν νερό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, είναι απόλυτα καθαρές, δεν έχουν εκπομπέ ούτε έχουν απόβλητα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστιες δυνατότητες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η ε, έρημη. Ε, η συντήρησή τους είναι πάρα πολύ εύκολη, διότι ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνει κανείς Ε, αποτελούν απλά συντήρηση των σχετικά απλών ε, τεχνολογιών που χρησιμοποιούν. Ε, επίσης, οι επιπτώσεις όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι ελάχιστες. Ε, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχει ε, πολύ γνώση στον τομέα αυτόν αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι όσο αποκτάει κανείς περισσότερες γνώσεις θα διαπιστώσει ότι η σκόνη ή η υγρασία ε, δεν δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις αυτές. Μπορεί να χτίσει κανείς αξιόπιστο σύστημα σχεδόν οπουδήποτε και ε, νομίζω ότι και μερικές ευρωπαϊκές χώρες το έχουν αποδείξει αυτό όσον αφορά την ανάπτυξη ε, μονάδων πολύ σημαντικό είναι ότι ε, ο χρόνος οικοδόμησης ε, είναι πολύ μικρός. Ε, μπορεί λοιπόν να δημιουργήσει κανείς τις εγκαταστάσεις αυτές με πολύ απλό τρόπο. πολύ σημαντικό είναι ότι μιλάμε για μονάδες, δηλαδή ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και κατά την συντήρηση και μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί και σε δόσεις μια τέτοια μονάδα να ξεκινήσει κανείς με 5, 10, 15 ΜΒ το ίδιο ισχύει και για τη συντήρηση. Μπορεί η συντήρηση να γίνει ε, σε κομμάτια. Επίση, δεν χρειάζονται σημαντικές ε, υποδομέ. Έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες για χώρου όπου δεν υπάρχει σήμερα υποδομή. Και τέλος μπορεί να το χτίσει κανεί αυτό οπουδήποτε. Φυσικά μπορεί να προτιμάει ε, ένας εργολάβο σε επίπεδη γη, αλλά και σε βουνοπλαγιά μια χαρά μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια μονάδα. μπορεί να μειωθεί και το κόστος ε, τη οικοδόμηση μια τέτοια μονάδα κατά 40%. Αυτό δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ε, υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης ε, το οποίο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για ερημικέ περιοχές. Οι ευκαιρίε που προσφέρουν ε, οι ηλιακές αυτές εγκαταστάσεις ε, είναι τεράστιες. Αυτή τη στιγμή ε, συνολικά στον κόσμο μπορεί να υπάρχουν 30.000 γιγαβάτ. Η χρηματοδότηση δεν είναι πια κάτι τελείως άγνωστο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα προσπαθήσω να σας κάνω γρήγορα την παρουσίασή μου ώστε να προλάβουμε να συζητήσουμε. Να σας δώσω μια εικόνα όταν μιλάμε για τεράστια έργα ε, φωτοβολταϊκά, μιλάμε συνήθως ε, για ε, μέγεθος 60-80 ΜΒ. Νομίζω ότι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, 290 ΜΒ στην Αριζόνα. Υπάρχει συμφωνία αγοράς ε, του ρεύματος ε, ε, από την PGEC στην Καλιφόρνια. Είναι λοιπόν πολύ ανταγωνιστικό το πρόγραμμα αυτό και μας δείχνει ότι περνάμε σε μια εποχή όπου τα προγράμματα αυτά γίνονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Κάτι που θέλουμε να πούμε εδώ είναι ότι η ηλιακή ενέργεια στις ερήμους έχει πολύ μεγάλη αξία είτε για τοπική κατανάλωση είτε για εξαγωγές. Ε, υπάρχει ανάγκη για τοπική κατανάλωση αλλά και η εξαγωγή είναι απαραίτητη για να γίνουν βιώσιμα τα ε, έργα αυτά. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, η φωτοβολταϊκή, γενικά η ηλιακή ενέργεια είναι ήδη σήμερα ανταγωνιστική επένδυση. Ε, ανανεώσιμη, ο ανανεώσιμος η, η, ε, ηλεκτρισμός ε, είναι ε, αυτό που βλέπετε. Θα συνεχίσουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αυτά, αυτές οι μονάδες ακόμα και μετά από 20 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν έτσι πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και σε περιοχές που σήμερα δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση. Τέλος, εμείς ε, ως ε, επιχείρηση αλλά και όλος ο τομέας έχουμε, λάβει, έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια ότι έχουμε ξεφύγει από τις ε, αγορές στήριξης, βρισκόμαστε στη μεταβατική περίοδο η οποία είναι κάπως δύσκολη. Και πρέπει να ξεπεράσουμε το στάδιο αυτό ώστε να γίνουμε μια βιώσιμη αγορά. Αυτό προσπαθεί να πετύχει αυτή τη στιγμή ο τομέας. Εάν ε, διπλασιάσουμε την κλίμακα, τότε ε, το κόστος ε, μειώνεται κατά 50%. Αυτός, αυτός είναι ο υπολογισμός που χρησιμοποιούμε εμείς και θα πρέπει να εξετάσει κανείς και τον κύκλο ζωής των προϊόντων, γιατί θέλει κανείς να χτίσει τα συστήματα αυτά με τρόπο βιώσιμο. Όταν Λοιπόν, ε, ε, ε, στήσει κανείς 7.000 τέτοια πάνελ, θα πρέπει να μπορεί να τα ανακυκλώσει μετά. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα σταθερό πολιτικό πλαίσιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπούλχαρτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Πολύ καλά μας παρουσιάσατε το θέμα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα λίγα λεφτά που έχουμε για τη συζήτηση νομίζω ότι πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Ό,τι έχει να κάνει με την ε, υποδομή θα το συζητήσουμε στη, ε, στη συνέχεια. Τρεις συναδελφοί έχουν ζητήσει το λόγο. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στα πολιτικά ερωτήματα και στο πρόγραμμα Desert Tech. Η κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θυμάμαι τους παλιούς καιρού τότε που προεδρεύατε. Τέλος πάντων. Πριν από οτιδήποτε άλλο, ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές, όλους τους εισηγητές, όλους τους προσκεκλημένους που ήρθαν και μας παρουσίασαν την δουλειά τους. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπαν και για τη Μεσόγειο, για τον Τεσερτέ κλπ. Τους ακούσαμε χωριστά τον καθένα, ο καθένα παρουσίασε το δικό του σχέδιο. Θα ήθελα όμως να του ακούσω και λιγάκι από κοινού μαζί. Τι εννοώ. Δηλαδή, πώς βλέπετε εσείς τη συνύπαρξη των προγραμμάτων, τι σχέση έχουν μεταξύ τους, Υπάρχει κάτι κοινό, υπάρχουν κάποιες συνδέσεις, κάποια συμπληρωματικότητα μεταξύ των προγραμμάτων σας. Αυτό θέλω να ξέρω. Ευχαριστούμε. Θα απαντήσετε μετά και Ο κύριος Τούρνες έχει τώρα το λόγο. Μία ερώτηση προς τον κύριο Κάουπ. Είπατε ότι τα δίκτυα μπορούν να ε, ε, υπάρξουν ε, μόνο αν έχουμε ε, διάφορες πηγές ενέργειας, όχι μόνο πράσινες, ε, αναφερθήκατε και στις γκρίζες και στις μαύρες. Ε, μαύρες πηγές ενέργειας δεν θέλω, διότι αυτό την εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από άνθρακα, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Επίσης θα ήθελα να τονίσω την ιδέα του κυρίου Στράους. Χρειαζόμαστε και την διάσταση, την εργασιακή για τους ανθρώπους στους τόπους αυτούς. Εσείς είσαστε παγκόσμιος παράγοντας. Τι πρέπει να γίνει ώστε να έχουμε παραγωγή στο Μαρόκο ή στην Τινησία ή στην Αίγυπτο. Ε, τι ακριβώς απαιτείται για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Τούρμες. Ο κύριος Ρίμπιχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Νίπλερ. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την ηλιακή ενέργεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, το κοινό ρυθμιστικό κέντρο στην Ιταλία που ε, κάνει ε, ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα τεστ, δοκιμές σε ηλιακά πάνελ. Ποιε θεωρείτε ότι είναι οι προκλήσει που συνδέονται με αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Πριν κάποιες μέρες ο Κλοντ Τούρμε σε συζήτηση με τον Επίτροπο Πίπαλξ που πριν ήταν ε, επίτροπος ε, για θέματα αναπτυξιακά η ενεργειακή πολιτική, ιδιαίτερα στην Αφρική και την Ασία, θα πρέπει ε, να τεθεί σε νέα βάση ε, και να δημιουργηθούν ε, περιφερειακές δομές που να μπορεί να στηρίξει την ευημερία και την παροχή ενέργειας στις χώρες αυτές. Έχετε δει κάτι τέτοιο, πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο έχει μέλλον και η τρίτη ερώτηση είναι όσον αφορά τον μηχανισμό ανάπτυξης. Κάποιες χώρες έχουν αποφασίσει να, ε, ε, την έξοδό τους από την πυρηνική ενέργεια. Πιστεύετε ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί έστω και εν μέρη να αντισταθμιστεί ε, στην Ευρώπη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρίμπιχ για την ερώτησή σας. Τέλος, ο Ιβο Μπέλετ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Αγγέλικα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που αργήσα. Ίσως να θέσω ερωτήσεις που ήδη να απαντήθηκαν από τους προσκεκλημένους μας, συζητώ και το προτέραν συγγνώμη. Σύντομα, για την σκοπιμότητα της, των εξαγωγών από τις χώρες της, της Νότιας Όχθης Μεσογείου προς την Ευρώπη και Τούμπαλιν. Πόσο σκόπιμο είναι κάτι τέτοιο, πόσο εφικτό είναι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς χάνεται πολύ ενέργεια. Πόσο λοιπόν είναι εφικτά όλα αυτά και έπειτα εσείς ε, από την Αμερική πού φτιάχνονται τα ισισορευτές στην Κίνα, στην Ένωση, στις ΗΠΑ υπάρχουν ε, δυνατότητες για παραγωγή είναι πολύ αργά. Τα έχουν ε, ήδη το μονοπόλιο, <laughs> αντές μην πω μονοπόλιο, αλλά πάση περιπτώσει τη μεγαλύτερη παραγωγή οι Κινέζοι. Ευχαριστώ κύριε Μπέλετ. Και εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πιστεύω ότι σημαντικό είναι για το πάνελ μας να ε, δούμε ε, τι θα θέλατε εσείς από εμά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε όλες τις επιθυμίες. Ε, κοιτώ και τον συνάδελφο του όσον αφορά την οδηγία ε, για τις ανανεμώσιμες πηγές ενέργειας ε, που υιοθετήθηκε το 2008. Συγκεκριμένη ερώτηση. Εάν εμείς πούμε ότι στηρίζουμε το όραμά σας, θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα. Τι, τι χρειάζεστε εσείς από εμά στην περίπτωση αυτή. Ε, θέλουμε να ε, ε, ε, καλέσουμε την Κομισιόν να φροντίσει για την γρήγορη εφαρμογή της οδηγίας στα κρατημέρια, αλλά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Θα πρότεινα τώρα ε, για τις απαντήσεις να ξεκινήσει ο κύριος Πούρχαρτ. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν σε εσά. Παρακαλώ κύριε Πούρχαρτ. Να προσπαθήσω να απαντήσω αντίστροφα με την ερώτηση για την Κίνα του κύριου Μπελέτ. Γιατί είναι μια αποσαφήνιση. Εμείς δεν παράγουμε στην Κίνα παράγουμε στη Γερμανία, στη Frankfurt Oder, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Στις ΙΠΑ έχουμε ένα εργοστάσιο στο Χάιο, στο Πάρισμπεργκ. Ήταν το πρώτο εργοστάσιο που φτιάξαμε και το δεύτερο που φτιάχνουμε στην Αριζόνα σε ένα μέρος που λέγεται μέσα. Έχουμε επίσης παραγωγή στη Μαλαισία και στο Βιετνάμ φτιάχνουμε ένα εργοστάσιο γιατί βλέπουμε ότι η ασιατική αγορά έχει απογειωθεί και πρέπει να είμαστε παρόντες. Και έχουμε επίση και ένα εργοστάσιο που το οποίο τώρα έχει παγώσει. Έχουμε ένα εργοστάσιο κάπου στη Γαλλία, γιατί δεν έχουμε αρκετή ορατότητα για την αγορά για να ολοκληρώσουμε αυτό το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζουμε από κοινού με την EVFF. Το πολύ σημαντικό θέμα είναι μέσω των συζητήσεων και στο Μαρόκο, το βασικό θέμα είναι η ορατότητα. Ορατότητα για μια αγορά, για επαρκεί όγκου που να επιτρέπουν οι κατασκευαστέ να έρθουν να επενδύσουν σε μια οποιαδήποτε χώρα, να... είτε είναι κατασκευαστέ, είτε είναι αν μπορέσουμε να, το, να τοποθετήσουμε επιτόπου ε, τους μηχανικούς, την, την κατασκευή, την παραγωγή, κερδίζει σε πάρα πολύ, ωφελείται και η χώρα, αλλά το σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο πολιτικής που επιτρέπει ορατότητα. Και ε, κάποιες από τις δυσκολίες που είχαμε στο παρελθόν, και φυσικά αυτό είναι και ζήτημα όταν είσαι σε μια διαδικασία όπου φτιάχνεις τα πράγματα ανά project, το πρόβλημα είναι ότι κάθε project το ίδιο μπορεί να δημιουργεί ορατότητα για αυτό το ίδιο, αλλά όχι για την αγορά στην οποία εγκαθίστασε. Ορατότητα στην Ευρώπη μέσω της εθνικής εφαρμογής της οδηγίας περί ανανεώσιμων και ένα πολύ θετικό παράδειγμα είναι η Γερμανία, για να έρθω μετά και στο γαλλικό παράδειγμα. Στη Γερμανία αποφάσισε πέρυσι να διπλασιάσει την αποδοτικότητα του εργοστασίου μας ε, και αυτό οφείλεται στο ότι η Γερμανία έδειξε μεγάλη σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να προχωρήσει με τα φωτοβολταϊκά. Για τον κύριο Ρούμπικ, να πω για το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα, είμαστε παδί του Ίσπρα του Κέντρου για τις Ανανεώσιμες και για την Ενέργεια κάνουν σπουδαίο έργο και μάλιστα όταν δει κανεί κάποιες από τις δοκιμές που έχουν κάνει για πρότυπα φωτοβολταϊκών και για ορισμένα πρότυπα ή, ε, μας έχουν βοηθήσει. Εμείς εγγυόμαστε 25 χρόνια, αλλά το κοινό ερευνητικό κέντρο εξετάζει 40 με 50 χρόνια. Αν δούμε λοιπόν ε, τη χρυσή εποχή της του ηλεκτρισμού, είναι τεράστια ευκαιρία αυτή και οι κυβερνήσει που έχουν μια ευφυή πολιτική για τι ανανεώσιμε θα το χρησιμοποιήσουν. Πέντε φορές μειώνεται το κόστος του ηλεκτρισμού, αν σκεφτεί κανείς πόσες γενιές θα το χρησιμοποιήσουν. Και είναι σημαντικό για ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιοχή, γιατί μιλάμε για βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Και από την άποψη της αναπτυξιακής πολιτικής επίσης είχαμε συζητήσεις με τον Πίπαλξ, και νομίζω και ο Μάικλ Όφεν θα πει κάτι γι' αυτό. Και ανέφερε και την κοινωνική συνιστόσα στην παρουσίασή μου. Η πρόσβαση απλά και μόνο στην ηλεκτρισμό δημιουργεί τεράστια ωφέλη όσον αφορά την παιδεία, την υγιεινή, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει βιομηχανία χωρί ηλεκτρισμό. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η πρόσβαση. Να συνδυαστεί η αναπτυξιακή πολιτική με την ενεργειακή είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση για τη Βόρεια Αφρική και για άλλα μέρη τη Μεσογείου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, για τις εξελίξεις για τον καθαρό μηχανισμό και την έξοδο από την πυρηνική ενέργεια της Γερμανίας και το δημοψήφισμα αυτό στην Ιταλία ως ένα θετικό σήμα για τις ανανεώσιμες, ναι. Να πω πως ναι, στη Γερμανία ήδη είδαμε ότι ο όγκος των φωτοβολταϊκών που έχει ήδη κατασκευαστεί έχει σταθεροποιήσει τους όρους, έχει σταθεροποιήσει τις συνθήκες. Είμαστε υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή με τη γερμανική κυβέρνηση για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι ανανεώσιμες στις απόδοση που γενικά χρειάζεται. Είναι βέβαια διαφορετικό γιατί είναι διαφορετικό το πώς χειρίζεσαι το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας όταν έχεις και την πυρηνική μέσα. Αλλά πάντως αυτό είναι και το θέμα με την, με τις, την οδηγία περί ανανεώσιμων, ότι οι ανανεώσιμες αποκτούν κεντρικό ρόλο. Νομίζω πως ναι, όσο και αν είναι ανταγωνιστικό το φυσικό αέριο για τις ανανεώσιμες, είναι το κατάλληλο συμπλήρωμα μαζί με την υδροηλεκτρική για να φτιάξεις γρήγορα και να είναι η βάση δηλαδή ανανεώσιμες και το φυσικό αέριο να είναι το τελικό συμπλήρωμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Στρός. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις ακούστηκαν. Κύριε Μαντουρέλ, επιμένετε στη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και σωστά. Οι επιδόσεις έδειξαν ότι έχουμε να κάνουμε με προγράμματα τα οποία είναι αρκετά διαφορετικά, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά δηλαδή μεταξύ τους. Το Desertec, γιατί δεν θα μιλήσω για τους άλλους, πρόκειται για βιομηχανικό με οικονομικούς ε, παράγοντες πρόγραμμα. Ενώ το ε, Solar Plan είναι περισσότερο πολιτικό, με αντίστοιχους στόχους βέβαια. Και όπως είπε και ο συνάδελφος από τη Solar, για να αναπτυχθούν όλα αυτά χρειάζεται ένα κατάλληλο και ευνοϊκό θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο. Ε, το συνεδεύτερο πρόγραμμα είναι πιο πολύ τεχνικής αρρωγής μέσων. Άρα λοιπόν τα προγράμματα αυτά δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, είναι συμπληρωματικά. Με προοπτικές διαφορετικές, με διαφορετική οπτική γωνία δηλαδή, αλλά είναι συμπληρωματικά και γι' αυτό και πρέπει να συνεργαζόμαστε και να επιδεικνύουμε κάθε φορά τη συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων μας. Οπότε δεν διαφωνώ καθόλου. Για αυτό που είπε ο Κλώτουρ Μέσο όσον αφορά την κοινωνική και βιομηχανική πολιτική στι χώρε νοτίω τη Μεσογείου και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ναι, επέμεινα και εγώ στην παρουσίασή μου γι' αυτό. Ότι δηλαδή. Τι λένε τα νούμερα. Υπάρχει μελέτη τη Παγκόσμια Τράπεζα που πρόσφατα είδε το φω τη ημέρα που δίνει μια τάξη μεγέθου και μιλάμε για 20 με 30% ε, για ε, δραστηριότητες ε, απασχόλησης. Στην Ισπανία, στις Πολιτείες φυσικά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η παραγωγή συστατικών πώς έχει. Ο χάλιβας είναι το πιο εύκολο για αυτούς. Αλλού χρειάζονται διαφορετικές τεχνολογίες. Υπάρχουν δύο εταιρείε στον κόσμο που φτιάχνουν ε, δέκτες. Πρέπει λοιπόν ή να αποφεληθούμε από την τοπική βιομηχανία στην Αίγυπτο, στο Μαρόκο ή και αλλού. Γίνεται, υπάρχει ήδη μια βιομηχανία παρούσα που μπορούν να παράγουν με αρκετή ποιότητα. Τώρα για τις ξένες επενδύσεις εξαρτάται από το μέγεθος της αγοράς, γιατί κάτω από ένα μέγεθος δεν έχει νόημα να παράγει κανείς τοπικά. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι να δούμε ποιες τοπικές επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να προχωρήσουν ε, με υπεργολαβία προς άλλους τομείς της βιομηχανίας. Έπειτα πρέπει να έχουμε και τις κατάλληλες πλατφόρμες, δηλαδή να υπάρχει σωστή επαγγελματική κατάρτιση, επιστημονική έρευνα κλπ. Τέτοιους μοχλούς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, κατά πόσο, λέει ο κύριος Μπέλτερ, όλα αυτά είναι εφικτά, λάβουμε υπόψη μας και την μεταφορά, Νομίζω πως ναι, το είπε και ο συνάδελφο. Οι συγκριτικέ μελέτες που λένε ότι ναι υπάρχει περισσότερο ήλιο στο νότο παρά στο βορρά εννοείται. Μας οδηγούν να πούμε πως ναι, εφόσον όμως έχουμε μια εταιρική σχέση από την οποία κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει όλε τι πτυχέ που θα την κάνουν να πετύχει στα ενεργειακά της προγράμματα και να είναι αποδοτική και το άρθρο 9 αποτελεί ένα στοιχείο μέσω το οποίο μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Συγχρόνως όμως πρέπει να αναπτύξουμε και την τοπική βιομηχανία και να διασφαλίσουμε μία παραγωγή κρίσιμης μάζας. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ναι. Τέλος για την ερώτηση της Πρόεδρου, που λέτε τι περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξακολουθεί να προβάλλει τα θέματα αυτά. Η ανάπτυξη που προστατεύει το περιβάλλον, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, αλλά και η αποκοινού ανάπτυξη των δύο όχθεων της Μεσογείου. Είναι και αυτό στρατηγική σημασία θέμα. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει όλα αυτά να τα προβάλλει. Να τα έχει δηλαδή ψηλά ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Να τα προβάλλει γιατί χρειάζεται αυτό. Και χρειάζεται επίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να έχουμε και αποτέλεσμα. Εμεί ξέρουμε ότι έχουμε το άρθρο 9. Εμείς έχουμε εντοπίσει ποια είναι τα μέσα που χρειάζονται αλλά χρειάζεται και πολιτική δουλειά και σε αυτήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο. Για μένα αυτά είναι τα σημαντικά, δηλαδή να ε, προβάλλεται πολιτικά το θέμα αυτό, να συζητιέται στην Ευρώπη αλλά και στις χώρες μέλη, ώστε όλοι να ε, διαθέσουν τα μέσα που χρειαζόμαστε για να πετύχει αυτό. Παρακαλώ, κύριε Στάρους. Ε, Η ερώτηση του Κλωτ ε, Τούρμε σχετικά με το πόσο μαύρο μπορούμε να κάνουμε το πράσινο ρεύμα. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σχετικά με έναν συμβιβασμό. Μηδόν ε, τόνους ε, διοξιδίου του άνθρακα αν θα εξέπεμπε μια μονάδα υψηλής απόδοσης. Εάν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε έναν μέσο όρο, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο. Η μεγαλύτερη μου επιθυμία και ήδη αναφέρθηκε από τον ιδιωτικό τομέα, θα... διότι ένα από τα βασικότερα εμπόδια είναι το κόστος της επένδυσης, ε, θα ήταν η καλύτερη διασφάλιση ε, κατά του κινδύνου, διότι 3 με 5% τόκι ή 12% για τη χρηματοδότηση μιας τέτοιας μονάδας ε, σχεδόν διπλασιάζει το κόστος παραγωγής. Καλύτερη ασφάλιση λοιπόν ε, απέναντι στους ε, κινδύνους θα ήταν επιθυμητό για τις ηλιακές εγκαταστάσεις. Ε, όσον αφορά το κόστος ε, μεταφοράς ε, και διανομής στην Ευρώπη, σας το έδειξα αυτό στην παρουσίασή μου. Όταν περάσουμε τις Άλπεις, για τον ε, καταναλωτή μπορεί αυτό να σημαίνει μείωση τελικά της ε, ε, θα, ήταν, θα είχαμε 10% ε, απώλειες, αλλά αυτό θα αντισταθμιζόταν από το ότι στον Νότο μπορούμε να παράγουμε ε, το διπλάσιο ρεύμα από ό,τι μπορούμε στις δικές μας χώρες. Έτσι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα δεν θα ήταν πολύ κακό τελικά. Ε, η οικονομικά είναι ελκυστικό το ρεύμα αυτό όταν φτάσει το ρεύμα στην Ευρώπη. Όχι στην Ισπανία, εκεί μπορεί να μην συμφέρει πολύ, αλλά πιο βόρεια. Ευχαριστώ κύριε Κάουπ. Ε, τέλος ο κύριος ε, Φανζόν. Οι περισσότερες ερωτήσεις ε, νομίζω ότι απαντήθηκαν επαρκώς. Ε, συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν από τους προλαλήσαντες. Δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η ερώτηση τι γίνεται με τα προγράμματα αυτά στη Βόρεια Αφρική. Ε, είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, μήπως ε, ε, μήπως ανταγωνίζονται υπερβολικά το ένα το άλλο. Εάν ε, χάναμε τώρα στο αρχικό στάδιο τόση ενέργεια στον ανταγωνισμό. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Προσπαθούμε να ε, δημιουργήσουμε τις μονάδες αυτές ε, με τρόπο παραπληρωματικό. Υπάρχει το ηλιακό σχέδιο για την Μεσόγειο και μαζί με, την, με τον πολιτικό τομέα και τις χώρες της Μεσογείου προσπαθούμε να αναπτύξουμε τα σχέδια αυτά. Η Desert όπως λέγεται το όνομα μόνο. Ε, είναι μια πρωτοβουλία ε, ε, που θέλει να προωθήσει ακριβώς το κίνημα αυτό, θέλει να επιταχύνει την δημιουργία μονάδων αυτών. Πολύ συχνά συνεργαζόμαστε σε ομάδες εργασίας, σε πάνελ κλπ. Είναι πολύ σημαντικό να ε, δημιουργηθεί αγορά όπου να μπορούν να επενδύσουν οι επιχειρήσεις μακροπρόθεσμα. Στη Γερμανία ξεκίνησε αυτό, τώρα σε 17 ε, οι επιχειρήσεις από 17 χώρες ε, λένε ότι θέλουμε να κοιτάξουμε και λίγο πέρα από τον δικό μας ορίζοντα. Όχι, δεν μιλάμε για τα επόμενα 5-10 χρόνια, μιλάμε για 40 χρόνια. Ε, σημαντικό είναι να δημιουργηθεί πλαίσιο στην Ευρώπη, στην ε, Βόρεια Αφρική, στην ε, Μέση Ανατολή, να υπάρξει σταθερότητα για τις μεγάλες επενδύσεις που χρειαζόμαστε, ώστε να έχουμε πέρασμα της ηλεκτρικής ενέργειας από, τις από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να έχουμε βιώσιμη ενέργεια. Επίσης σημαντικό είναι ότι ο τομέας ε, λέει να κοιτάξουμε πέρα από τον δικό μας ορίζοντα, να μην ε, κοιτάξουμε μόνο τι θέσεις εργασίας, εργασίας δημιουργούνται στις δικές μας χώρες, ε, αλλά τι θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και σε άλλες χώρες παραγωγής και με τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Φροντίζουμε λοιπόν τα προγράμματά μας ε, να συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Υπάρχει η γαλλική πρωτοβουλία NetQuit ε, που ασχολείται με το θέμα του δικτύου. Όλα αυτά ταιριάζουν πολύ καλά το ένα με το άλλο. Κατά τη γνώμη μου η Desertec ε, συνεχίζει να είναι κάπως μοναδική διότι ασχολούμαστε με την πολύ μακροπρόθεσμη προοπτική για τα επόμενα 40 χρόνια Ε, ενώ η ΜΕΝΤΕΜΙΠ κοιτάει τα επόμενα 10 με 15 χρόνια, είμαι, σίγουρη, είμαι σίγουρος όμως ότι ε, θα κοιτάξουν και πιο μακροπρόθεσμα. Επίσης, ο Κλωτ Τούρμες ε, έθεσε ένα θέμα. φυσικά, στόχος μας δεν είναι να ενισχύσουμε την πυρηνική ενέργεια ή την ενέργεια από, ορυκτές, από ορυκτά καύσιμα. Θέλουμε ε, η υποδομή του δικτύου να εξυπηρετεί ε, κυρίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κύριος Ρούπιχ έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με την βιωσιμότητα των ε, εξαγωγών ηλιακής ενέργειας. Η μακροπρόθεσμη προοπτική μεταφορά σε, μεγάλα, σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα αναπτυχθεί η αγορά στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αφρική, καθώς και στη Μέση Ανατολή. Ποιες ε, θα είναι οι δυνατότητες ε, και ποια θα είναι η διαμόρφωση των τιμών. Το να μεταφέρουμε ρεύμα από ένα σημείο α προς ένα σημείο β θα γίνει μόνο εφόσον οι τιμές είναι ενδιαφέρουσες. Ε, δεν θα ε, θα επενδύσουμε σε ένα δίκτυο μόνο εφόσον η διαμόρφωση των τιμών το ε, δικαιολογούν αυτό ε, μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη των τιμών στους διάφορους τομείς της αγοράς και θα πούμε τότε ότι μόνο τότε έχει νόημα να επενδύσουμε σε κάποια μέρη του δικτύου, κάποια κομμάτια του δικτύου. Επίσης, ε, μας ρωτήσατε ποιος είναι ο κατάλογος των επιθυμιών μας. Ε, θέλουμε ε, ο Άγιος Βασίλης να μας φέρει όλα όσα θέλουμε. Η δική μου μεγαλύτερη επιθυμία θα ήταν η Ευρώπη μαζί με την Βόρεια Αφρική να καταλάβουν ότι μακροπρόθεσμα έχουμε πολύ λίγες επιλογές όσον αφορά την ενέργεια. Έχουμε την υδροελεκτρική ενέργεια, την αιωλική, τη βιομάζα και έχουμε και κάποιες άλλες επιλογές. Δεν είναι όμως πολύ μεγάλες οι πηγές αυτές. Στην Βόρεια Αφρική και στην Μέση Ανατολή υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες η αεολική και η ηλιακή ενέργεια. Και στο πλαίσιο και θέλουμε να δημιουργηθεί ένα ε, σταθερό πλαίσιο Θα πρέπει λοιπόν σε συνεργασία με τον τομέα και τους απαραίτητους φορούς την τεχνολογία που γνωρίζουμε ε, να την ε, εισάγουμε στις αγορές. Και έτσι ε, φτάνω και στο θέμα που αναφέρθηκε φυσικά. Ε, συμφωνώ με τον Άλπρεχτ Κάουπ, όπως και με μικρά παιδιά, όταν μπορούν μόνα τους να σταθούν στα πόδια τους, ε, θα πρέπει να τους δώσουμε την αυτονομία τους. Το ίδιο ισχύει και για ε, τα φωτοβολταϊκά στη Βόρεια Αφρική. Βρίσκονται σε καλό δρόμο και πολύ γρήγορες είναι οι εξελίξεις. Το βλέπουμε αυτό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τιμές πέφτουν, ε, η ποιότητα είναι εξαιρετική. Όλα αυτά πηγαίνουν λοιπόν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και την έχουμε το προβληματικό μας παιδί, ε, την ε, ηλιοθερμική ενέργεια. Αυτή έχει μακροπρόθεσμα, μεγάλες δυνατότητες, μπορεί να αποθηκεύσει κανείς την ε, ενέργεια. Είναι σήμερα όμως προβληματικό παιδί. Ε, όλα, ε, ε, το, το, προβληματικό παιδί αυτό όμως θα απαιτήσει κάποια χρήματα μέχρι να σταθεί στα πόδια του. Θα χρειαστούμε λοιπόν την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα χρειαστούμε επίσης την συνεχιζόμενη εφαρμογή του άρθρου 9. Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τρόποι υλοποίησης εφαρμογής του άρθρου 9. Δεν ξέρω σε τι βαθμό υπάρχει εναρμόνιση στην Ευρώπη. Δεν ξέρω καν αν επιτρέπεται να λέω τη λέξη αυτή εδώ πέρα. Πάντα πρέπει να προσέχει κανείς. Ε, θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα πιλωτικά προγράμματα και θα πρέπει να τονίσουμε την ολοκλήρωση της ε, αγοράς. Θα χρειαστούμε μια γενική συμφωνία ανάμεσα στην Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ε, έναν ενεργειακό χάρτη. Το ξέρετε αυτό από τη δεκαετία του 80. Ε, θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή σταθερό πλαίσιο. Έτσι θα έχουμε τη βάση, θα έχουμε τις συνθήκες πλαίσιο για ε, την ενεργειακή αγορά. και θα πρέπει να ε, παρακολουθήσετε τις εξελίξεις αυτές και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ε, να υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας ε, να υπά... και στον τομέα της εκπαίδευσης να γίνονται ανταλλαγές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει το Desert Tech University Network, το δίκτυο πανεπιστημίων. Αυτό δεν θα πρέπει να το υποτιμήσουμε. Σε όλες αυτές τις χώρες, αλλά και στην Ευρώπη, Υπάρχει πολλή τεχνογνωσία και νέοι άνθρωποι ασχολούνται με, ε, ε, την ανάπτυξη του τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την ε, συζήτηση αυτή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ομιλητές ε, και χωρίς καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συνάδελφο Ριέρα Μαντουρέλε για να ηγηθεί των συζητήσεων στο επόμενο πάνελ. Ευχαριστώ. Bueno, buenas tardes. Vamos pues a comenzar Καλησπέρα και από μένα. Περνάμε στο επόμενο πάνελ, το δεύτερο πάνελ. Θα μιλήσουμε για τα δίκτυα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρειάζονται ισχυρά, δυνατά δίκτυα και όπως το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας, αλλά ανέφεραν και κάποιοι από τους προσκεκλισμένους μας μέχρι τώρα, υπάρχουν διάφορες κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε αλλά και να ξανασχεδιάσουμε ενδεχομένω δίκτυα ηλεκτρισμού στην νότια πλευρά της Μεσεγείου για να ανταποκρίνονται και σε προδιαγραφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειες, ώστε αυτές οι τελευταίες να καλύψουν μεγάλο μέρος των αναγκών των χωρών αυτών. Έπειτα χρειάζεται διασύνδεση μεταξύ των ίδιων των χωρών οτίως της Μεσογείου. Να μην υπάρχει ο σημερινός κατακαιρματισμός και να υπάρξει έτσι μια ισχυρή περιφέρεια. Άρα πρέπει να επενδύσουμε στην διασύνδεση μεταξύ των ε, δύο πλευρών της Μεσογείου, ώστε όπως είπε και ο κύριος Τούρμες, η ενέργεια που μεταφέρεται να είναι από πηγές ανανεώσιμες. Πρέπει να φροντίσουμε επίσης και τη διασύνδεση με ταξί της νότιας πλευράς της Μεσογείου και της Ευρώπης, τόσο της νότιας όσο και του βορρά. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο στραγγαλισμός όπως υπάρχει σήμερα στα σύνορα Ισπανίας-Γαλλίας. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά έχουμε τρει εξαίρετους ομιλητές. Έχουμε πρώτα απ' όλα εξ αριστερών μου τον κύριο Ζορ Ντεμον Μοντραβέλ που είναι Γενικός διευθυντή της MedGrid ο οποίο θα μας ε, αναφέρει τους στόχους που έχουν ε, για να φτιάξουν αυτό το super grid που συνδέεται στις δύο πλευρές της Μεσογείου. Μετά έχουμε τον κύριο Χουάν Μανουέλ Ροντρίγκε, που είναι εκπρόσωπος του Red Electrica και υπεύθυνο ε, διεθνών οργανισμών. Σίγουρα και αυτός έχει να μας μεταφέρει πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία γιατί η Electrica είναι ο διαχειριστής ο οποίος έχει πάει πιο μακριά όσον αφορά την ε, συμπερίληψη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυό τους. η Desertec και το Red Electrica έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την Ισπανία προκειμένου να φέρνει ενέργεια από τη Βόρεια Αφρική. Έπειτα έχουμε και τον κύριο Μαβοήλ Ναβράνη από το Μαρόκο στην άλλη μεριά, ο οποίος θα μας μιλήσει και για τα δύο προηγούμενα προγράμματα. Το Μαρόκο αποφάσισε να στοιχηματίσει σε ίδιους πόρους και να πετύχει το στόχο 42% ανανόσιμες πηγές ενέργειας για το 2020. Ο κύριος Σαμαρανέ, ο οποίος είναι μέλος του ε, Συμβουλίου του Μαρόκου για την ηλιακή ενέργεια, θα μας εξηγήσει τις προσπάθειες που κάνει η χώρα του για να πετύχει το στόχο αυτό. Και θα μας μιλήσει επίσης και για την ε, σχέση του Μαρόκου με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να έχουμε ανανόσιμες πηγές ενέργειας εκατέρωθεν της Μεσογείου. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους εισηγητές και θα ξεκινήσουμε με την ανάποδη σειρά. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μίτα Γάμετ πρώτα απ' όλα, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου του Μαρόκο για την ηλιακή ενέργεια. Έχετε το λόγο. Merci, Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ όπως και οι προηγούμενοι μιλητές να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ρόλ που μας έδωσε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο το μαροκινό ηλιακό πρόγραμμα και να μοιραστούμε μαζί σας τους προβληματισμούς μας ε, καθώς και τις εργασίες που κάνουμε μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 9. Καταρχήν θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για να αντιληφθείτε το πλαίσιο. Ήδη συζητήθηκαν κάποια πράγματα. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα προσωπικά να επιμείνω σε κάποιες λέξεις κλειδιά που αναφέρθηκαν. Ακούσαμε στο προηγούμενο πάνελ, το κόστος ε, ανάπτυξης, την ορατότητα, την ευημερία και την γυτνίαση. Είναι όλα αυτά στοιχεία κλειδιά που καθορίζουν τα προγράμματα για τα οποία μιλάμε. Πέρα δηλαδή από προγράμματα είναι ένα όραμα. Εξαρτάται από το σημείο αφαίρεσης στο οποίο βρισκόμαστε, από το ύψος ε, από το οποίο προσεγγίζουμε αυτά τα προγράμματα, την οπτική γωνία. Βασικά όμως συζητάμε για την ενέργεια της τρίτης χιλιετίας, μιλάμε για αλλαγή ε, παραδειγμάτων ή προτύπων. Και σε σχέση με αυτά θα πρέπει να μετρήσουμε τη σημασία των ε, εργασιών. Και γι' αυτό επέμεινα για τη σημασία της σημερινής παρέμβασης και τη τιμή που μου κάνετε να συμμετέχω σε αυτές τις εργασίες το Μαρόκο. Είναι μια νέα χώρα. Ε, μια χώρα όπου ο πληθυσμός, ε, πάνω από το 60% του πληθυσμού είναι κάτω των 35 ετών. Είναι νέο λοιπόν ε, με, όσον αφορά την ανάπτυξή της που πρέπει να τροφοδοτηθεί από την ενέργεια την ανάπτυξη της ενέργειας. Οι ανάγκες ενέργειας του Μαρόκου θα διπλασιαστούν μέχρι το 2020 <coughs> και μέχρι το 2030 θα ξαναδιπλασιαστούν, θα τετραπλασιαστούν δηλαδή ανάμεσα στο σήμερα και το 2030. Τι σημαίνει αυτό, καταλαβαίνετε ποια σημασία έχουν οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν. Σας δίνει τη δέσμευση στην οποία την οποία είμαστε ε, ε, ε, αναγκασμένοι να αναλάβουμε όταν μια χώρα που εδώ και πάνω από μια δεκαετία γνωρίζει ανάπτυξη της τάξης του 5% και που αυτή η ανάπτυξη εντάσσεται σε μια δυναμική επιτάχυνσης. Όλοι θα θυμάστε την πρόσφατη επικαιρότητα, άρα όλοι μας θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις ε, προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και να τις διατηρήσουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στηριχθούν περισσότερο τα τομεακά προγράμματα για να εξασφαλιστεί η απασχόληση όλες αυτής της νεότητες ο ηλεκτρισμός και η ενέργεια γενικότερα αποτελούν ένα σημαντικό βασικό στοιχείο αυτής της αναζήτησης στήριξης της ανάπτυξης. Είμαστε μια χώρα που εξαρτάται κατά πάνω από το 90% για να πω από το 97% από τις, την ορυκτή ενέργεια την οποία εισάγουμε από το εξωτερικό. Όσον αφορά αυτά τα δύο στοιχεία, να τα εξισώσουμε, αποδεικνύεται απλούστατα και τάχιστα πως αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί μέσω ακόμα και βράχη πρόθεσμα. Ξεκινώντας με αυτό το στοιχείο λοιπόν, αλλά και με βάση την βούληση που εκφράζεται στο ε, ανώτατο ε, κρατικό επίπεδο, μια βούληση να, να, να έχουμε μια οπτική για βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μια επιλογή που γίνεται μέσα στο πλαίσιο μιας ε, ανάπτυξης, γιατί σήμερα δεν υποχρεωνόμαστε εμείς να περιορίσουμε, ως Μαρόκο να περιορίσουμε τις εκπομπές ρήπων, του θερμοκηπίου, εμείς ε, ε, ηθελημένα ακολουθούμε την πράσινη ανάπτυξη ώστε να αποφύγουμε οι νέες γενιές να χρειάζεται να επανέλθουν για να διορθώσουν ε, τις, τα λάθη το, τα δικά μας. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτή τη διπλή προσέγγιση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πλέον η μοίρα μας, ας το πούμε έτσι, αλλά και η λύση που επί της οποίας ε, θα πρέπει να εγγύψουμε. À partir de là, les autorités marocaines se sont fixées des objectifs. Οπότε, με βάση αυτά τα στοιχεία, οι ε, μαροκινές αρχές έθεσαν στόχους έτσι ώστε μέχρι το 2020 να έχουν φτιάξει ενεργειακή απόδοση ε, μέχρι και 42% της ε, ισχύω ε, το... Ε, για τη χώρα μας. Έχουμε, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε δηλαδή ηλιακή ενέργεια, αιωλική και υδροηλεκτρική. Για να σας δώσω το μέτρο τώρα όλων αυτών. Η ηλιακή ενέργεια αυτή τη στιγμή δυστυχεί πάνω από το, σε πάνω από το 30%. Καταλαβαίνετε ποια είναι η δέσμευσή μας, ε, εφόσον πρόκειται για αναπτυσσόμενη χώρα ε, τη της Βόρειας Αφρικής. Εάν το καταφέρουμε αυτό θα έχουμε κάνει οικονομία εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 3,7 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Διόλου αμεληταία οικονομία λοιπόν. Τώρα μπορεί κανείς να μιλήσει αν θα είναι η ηλιακή ενέργεια, η αιωλική κτλ. Μα η ασφάλεια βρίσκεται στη διαφοροποίηση. Εδώ είναι ένα θέμα στρατηγικό, επί του οποίου η διαφοροποίηση είναι το ζητούμενο. Για να φτιάξουμε αυτή την στρατηγική, το Μαρόκο έχει φτιάξει ένα ολόκληρο πλωστάσιο κινήτρων με σαφές νομοθετικό πλαίσιο μέσω της οδηγίας για την ε, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε φιλελεύθερη χώρα, Θα ενθαρρύνουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουμε ήδη πειραματιστεί με την ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρισμού που αντιπροσωπεύει ένα δύο λαμελιτέο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται στο Μαρόκο. Ε, επίσης έχουμε και την, ναι, τη, διανομή, είναι κάτι το οποίο γίνεται ούτως ή άλλως περιφερειακά και έχουμε ενθαρρύνει και την αυτοπαραγωγή. Την ίδια παραγωγή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Έχουμε δημιουργήσει ένα θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για να υλοποιηθεί αυτός ο βασικός στόχος που είναι να, να οδηγηθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αποτελέσουν αυτές ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα μας. Το πρόγραμμα το ηλιακό εντάσσεται μέσα σε μια ολοκληρωμένη εικόνα και με πολλές διαστάσεις, με προοπτικές περιφερειακής ολοκλήρωσης. Μιλάμε για αξιοποίηση των φυσικών πόρων, το ανανεώσιμο αυτού πόρου, αλλά και όσα στρέφονται γύρω από την δημιουργία βιομηχανικών θυγατρικών ανταγωνιστικών, δηλαδή κατάρτιση, έρευνα και ανάπτυξη, ε, βιομηχανική ολοκλήρωση. Έχουμε δεσμευθεί να φτιάξουμε 2.000 ΜΒ ηλιακής ενέργειας για την τοπική μας κατανάλωση. Αν σήμερα το Μαρόκ δεν υλοποιήσει μέχρι το 2020 τα 2.000 ΜΒ, ο δημόσιος φορέας θα πρέπει να αντικαταστήσει αυτά τα 2.000 ΜΒ με τον άνθρακα, με παραγωγή από άνθρακα, γιατί θα μας λείπουν τα 2.000 αυτά ΜΒ. Άρα λοιπόν το Μαρόκο υλοποιώντας αυτό το πρόγραμμα δίνει ορατότητα και στις άλλες πρωτοβουλίες, στις περιφερειακές, είτε είναι αυτές πολιτικές, είτε είναι βιομηχανικές και δεσμεύεται πλήρως σε αυτό το επίπεδο. Είναι δηλαδή ένα άνοιγμα που όμως χρειάζεται και πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Το άρθρο 9, εμείς στο Μαρόκο Χαιρόμαστε για αυτή τη διάταξη και ευχαριστούμε τα μέλη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, διότι αποτελεί μια απάντηση στις ε, ε, περιβαλλοντικές ε, και ενεργειακές φιλοδοξίες της Ευρώπης, αλλά μπορεί να αποτελέσει έναν μοχλό για μια αμοιβαία ωφέλιμη συνεργασία. Ταυτόχρονα βέβαια δεν πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα καλύψει όλες τις ανάγκες της Μεσογείου. Πρέπει να, χρειαζό... να έχουμε μηχανισμούς που να είναι στο ύψος των προσδοκιών, των φιλοδοξιών, οι οποίες είναι πολύ ψηλές. Πριν από λίγο γίνει λόγος για τον Άι Βασίλη. Ε, τι να προλάβει ο Άι Βασίλης, είναι μακρύς ο κατάλογος. Θα μπορούσαμε ωστόσο να πούμε ότι είναι και μικρός. Γιατί δεν λείπουν τα κεφάλαια ο αγοραστής της, του ηλεκτρισμού είναι που λείπει. Και θα πρέπει να αγοράσει με έξυπνο τρόπο. Η ιδέα αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλλει στις διώχτες της, της ε, Μεσογείου ε, στην αλλαγή των προτύπων. Πρέπει να κάνουμε μια απόδειξη βέβαια, μια επίδειξη μάλλον το ο Μαρόκο υλοποιεί το πρόγραμμα WERZAZAD, επενδύει σε αυτό και είναι μια επίδειξη για το ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αποδοτικές, μπορούν να κινητοποιήσουν χρηματοδότηση, μπορούν να παράγουν καθαρό ηλεκτρισμό, αλλά και είναι και προβλέψιμες. Δηλαδή μπορείς να αποθηκεύσεις, πράγμα που επιτρέπει να ενταχθεί στα δίκτυα με ήρεμο και νυφάλιο τρόπο. Αλλά γιατί το στόχος είναι να φτάσει αυτή ο ηλεκτρισμός σε ίδιο επίπεδο με τις ορυκτές ενέργειες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια αγορά, μια αγορά ώστε οι βιομηχανίες, να, οι βιομηχανοί μάλλον μπορούν να επενδύσουν, να μπορούν να αυξήσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες. Και άρα χρειάζεται ορατότητα και δέσμευση μακροπρόθεσμη για να μπορέσουν οι ηλιακές ενέργειες να είναι οι ενέργειες του μέλλοντος αν χρειαζόταν να σκάσουμε ένα βεγγαλικό, δεν θα χρησιμεύσει τίποτα για τη δημιουργία μιας ε, ε, ολόκληρης, ε, ενός ολόκληρου κλάδου. Πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, σχέδιο που να εγγυάται την βιωσιμότητα βιωσιμότητα λοιπόν από το πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξασφάλιση και για παγίωση των ε, ε, παροχών των συνεργασιών. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το, τα κεφάλαια που πρέπει αρχικά να καταβληθούν, είναι το, η απόδοση αυτών των κεφαλαίων, η απόσβεσή τους. Δηλαδή, μπορεί η τιμή του ισκυλοβατόρα από τις ηλιακέ ενέργειες να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 35% τη τιμή τη παραδοσιακή ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει όμως να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να δείχνουμε, να αποδεικνύουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οι προσπάθειες ε, θα πρέπει τώρα να γίνουν στο μέγιστο βαθμό για να στηριχθεί αυτό το παιδάκι που δεν είναι άρρωστο, είναι απλώς μικρό και αναπτύσσεται. Χρειάζεται πολύ προσοχή και πολλές ώρες αφουσίωσης, ώστε να γίνει παιδί, μετά έφηβος, μετά ένας έφηβος ε, πιο όριμος που θα, και ένας νέος που θα μπορεί να δουλέψει μόνος του και να σταθεί μόνος του. Χρειάζονται λοιπόν μηχανισμοί συμβάσεων, μια αγορά ηλιακής ε, ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως να εξελιχθεί και το άρθρο 9. Θα πρέπει δηλαδή να εξελιχθεί το άρθρο 9 περνώντας από την προαίρεση στην υποχρέωση. Γιατί σήμερα αυτό που λέει η οδηγία είναι ότι οι χώρες που δεν έχουν ε, τηρήσει τις δεσμεύσεις τους μπορούν να ανατρέξουν σε εισαγωγές. Να καταφύγουν σε εισαγωγές. Αλλά και στο τελειότερο κόσμο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πως αυτή η δυνατότητα, αυτή η επιλογή θα μπορούσε να μετατραπεί σε υποχρέωση που να λέει απλά αφού έτσι και λίγο στον Άι Βασίλη τα λέμε μα Άι Βασίλη κάνε το θαύμα σου και κάνε έτσι ώστε η, το κομμάτι της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη-μέλη το 0,5% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από τις νότιες χώρες. Κάτι τέτοιο είναι απόλυτα εφικτό. Εφικτό στο πλαίσιο της σημερινής εκδοχής ε, της, ε, σύστασης, της, της σύνταξης οδηγίας για τα πιλωτικά προγράμματα, αλλά για να περάσουμε στο αύριο σε μια χώρα που θα στηρίξει ολόκληρη βιομηχανία πρέπει να ανατρέξουμε σε μέσα βιομηχανικά. Θα πρέπει αυτή η εξέλιξη να γίνει χωρίς περίπλοκες ιστορίες, μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει ήδη. Τα στοιχεία αυτά να καταστούν ε, πάνω κάτω υποχρεωτικά για την πρώτη φάση και αυτή η συμβολή που φαίνεται εμένα ότι είναι ελάχιστη να δώσει ορατότητα για τους ε, φορείς και να δημιουργήσει την ε, απαραίτητη όθηση. Εμείς καλούμε την Κομισιόν να έρθει να επισκεφτεί την, ε, το Μαρόκο, να, να δείξουμε ακριβώς πόσο ε, είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες στο Μαρόκο, γιατί τέτοια κοινά προγράμματα δημιουργούν αξία για όλους τους συμμετέχοντες. Και να δούμε αύριο μεθαύριο τι θα έχει φέρει ο Άγιος Βασίλης ε, στο τζάκι για τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προπτική αυτή που μας δώσατε. Ξέχασα να σας πω ότι είχαμε προβλέψει το πολύ για 10 λεπτά να μιλήσει ο καθένας από τους ομιλητές και ίσως ε, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι πρέπει να τηρείτε το χρόνο σας. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μονταβέλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να σας παρουσιάσω το Metacrit. γύρω από τη Μεσόγειο. Επιμένω για το ότι πρόκειται για κάτι που θέλουμε εμείς να εφαρμόσουμε, όχι κεντρικά από το Παρίσι, αλλά θέλουμε πρώτα να έχουμε ένα όραμα και μετά να προχωρήσουμε σε συνεργασία με όλες τις χώρες που βρίσκονται γύρω από τη λεκάνη της ε, Μεσογείου. Ο κύριος Στρός υπενθύμησε λίγο το ιστορικό υπόβαθρο, πάντως πρέπει να ξέρετε ότι το MedGrid είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα ηλιακής ενέργειας. Ακόμα και αν το πεθύμιζε και ο κύριος τώρα, το λέω και εγώ, ότι προβλέπουμε την ε, επιπλέον χωρητικότητα 20 ΜΒ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 20 ΓΒ λοιπόν, ε, και από τις δύο πλευρές ε, της Μεσογείου. Και αυτό για το 2020. Βέβαια, μπορεί να καταλήξουμε να έχουμε ακόμα περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Αλλά στην αρχή ήμασταν σκεπτικοί ακόμα και για αυτό το στόχο. Τώρα εννοείται ότι η οικοδόμηση αυτή νέας χωρητικότητας θα ικανοποιήσει τις τοπικές ανάγκες. Ο κ. Σαμουράν υπενθύμησε πριν ότι η κατανάλωση ενέργειας στο Μαρόκο θα διπλασιαστεί μέχρι το 2020. Άρα πρέπει να ικανοποιηθούν πρώτα οι τοπικές ανάγκες, η τοπική ζήτηση αλλά μετά πρέπει να δούμε και την εξαγωγή προς την Ευρώπη. Προς το παρόν, σε σχέση με αυτά τα 20 ε, γιγαβάτ, προβλέπουμε 5.000 μεγαβάτ να εξάγονται προς την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια εξέλιξη και στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας γύρω από τη Μεσόγειο. Και όχι μόνο εξαιτίας της ανάπτυξης ε, παραγωγής εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αλλά και για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες κατανάλωσης λόγω της ανάπτυξης. Το MedGrid λοιπόν θα λάβει υπόψη όλα τα σχέδια παραγωγής και τα μελλοντικά και όχι μόνο για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και για όλες τις πηγές. Γιατί τώρα χρειάζεται η εξέλιξη αυτή στα δίκτυα μεταφοράς, πρώτα απ' όλα γιατί πρέπει να υπάρχει μια ολοκλήρωση του δικτύου. Δεύτερον, να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού, γιατί αν ενισχύσουμε το δίκτυο, ενισχύουμε και τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις χώρες νοτίως της Μεσογείου με τις χώρες βορείως της Μεσογείου και γιατί θέλουν και μια ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρισμού στην λεκάνη της Μεσογείου. Υπενθυμίζω μάλιστα ότι ακριβώς αυτή είναι και η διαδικασία που αναπτύχθηκε όταν δημιουργήθηκαν και τα πρώτα δίκτυα ηλεκτρισμού στην Ευρώπη με αλληλεγγύη μεταξύ των συστημάτων και τα τελευταία χρόνια με μια εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού. Τι ακριβώς είναι το Medgrid? Είναι μια βιομηχανική πρωτοβουλία, όπως και η Desert για παράδειγμα. Περιλαμβάνουμε 21 επιχειρήσεις, 20 μετόχους και έναν στρατηγικό εταίρο. Ορισμένοι έρχονται από τις χώρες νοτιούς της Μεσογείου, θα πάνε αργότερα σε αυτό. Είναι μια επιχειρήση πολύ νέα. Τον Ιανουάριο του 2011 επίσημα άρχισε να λειτουργεί και η έδρα μας είναι στο Παρίσι. Θα σας πω δύο λόγια τώρα για τους εταίρους μας. Θα ξεκινήσω από αυτούς του Νότου. Έλεγα ότι το MedGrid είναι ένα πρόγραμμα από κοινού ανάπτυξη. Γι' αυτό και προσπαθούμε να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερου εταίρου από τι νότιε χώρε. Ο πρώτο είναι το Μαρόκο. Το η Εθνική Επιχείρηση Ενέργειας, μετά από το Κατάρ, ε, Συρία, ε, η το Πανμέντ. Και μεταξύ των πιο ευρωπαϊκών εταίρων θα αναφερά διαχειριστές δικτύων όπως είναι η Ερελέκτρικα, όπως είναι η ΕΡΤΕ, η ΤΕΑ στην Ιταλία η Άστομα, οι η ΕΝΕΞΑΝΣ και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας όπως είναι η ΕΝΚΟΑ ή η ΣΟΙΤΕΚ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η MedGrid αναπτύσσοντας το δίκτυό της. Πρώτα απ' όλα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των ε, εγκαταστάσεων και μας επιτρέπει και ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών της Μεσογείου, αλλά και ε, μέσα στην Ευρώπη, βάσει το άρθρο 9, στο οποίο αναφερθήκαμε τόσο πολύ. Έπειτα υπάρχει μια ασφάλεια εφοδιασμού με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι επιτρέπονται εισαγωγές, εξαγωγές και ανταλλαγές προς τις δύο κατευθύνσεις. Μιλάμε για εξαγωγή από τον νότο προς το βορρά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ ε, συστημάτων ηλεκτρισμού είναι κάτι που δουλεύει αμφίδρομα. Την απόδοση θα την έχουμε στο μέγιστο εφόσον υπάρχουν ε, ανταλλαγές προς τις δύο κατευθύνσεις, αφίδρομες. Ποιοι είναι τώρα οι πέντε στόχοι του Medgrid. Πρώτον, θέλουμε να καθορίσουμε ε, το σχέδιο των δικτύων γύρω από την ε, Μεσόγειο και μέσα από τη Μεσόγειο και αυτά εν ώψη του 2020-2025. Αυτό το σχέδιο, το σχήμα, λαμβάνει υπόψη όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τις ανώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και άλλες μορφές, μια που πρόκειται για την ανάπτυξη της παραγωγής. Δεύτερον, θέλουμε πρόθεση ενός θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου με εναρμόνιση. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό και νωρίτερα. Πάντως, στην αρχή της δημιουργίας του δικτύου ηλεκτρισμού στην Ευρώπη χρειάστηκε να καθοριστούν κανόνες για να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές, πώς θα αμείβεται το transit, οι χώρες δηλαδή από όπου περνάει ε, το ηλεκτρικό ρεύμα. Ε, όλοι αυτοί οι κανόνες υπάρχουν γύρω από τη Μεσόγειο. Υπάρχει αναρμόνιση. Τρίτον, αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεων που γίνονται στα δίκτυα υποδομών. Γιατί αν θέλουμε να προσελκύσουμε επενδυτές πρέπει να τους αποδείξουμε ότι αποδίδουν οι επενδύσεις τους. Θέλουμε επίση να αναπτύξουμε συνεργασίε σε τεχνικό και τεχνολογικό επίπεδο μεταξύ, και, ε, ε, νότου και ανατολικών χωρών. Με όλους τους εταίρους μας. Και τέλο θέλουμε να προωθήσουμε τεχνικές συνεχού συνεχούς ρεύματος υψηλής Γιατί ξέρετε εδώ πρόκειται για μεγάλες αποστάσεις, υποθαλάσσια κυρίως, είναι τεχνικές συνεχούς ρεύματος που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Και θα τελειώσω με δύο λόγια για την Tech Industrial Initiative. Ποιο ρωτήσατε εσεί, κύριε Πρόεδρε κάτι για τη συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων αυτών. Και συχνά το MedGrid το παρουσιάζουμε σαν ένα πρόγραμμα που ανταγωνίζεται το άλλο. Όχι. Είναι δύο συμπληρωματικά προγράμματα. Εξάλλου θα υπογράψουμε και συμφωνίε συνεργασία. Και για να σα τα πω όλα, χρόνο δεν είχαμε, επειδή οι υπουργοί έχουν πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και θέλουν όμω να είναι παρόντε στην υπογραφή αυτή τη συμφωνία. Κάτι πολύ σημαντικό και για τι δύο επιχειρήσει είναι μια συνεργασία που επιθυμούμε να είναι μακρά και καρποφόρα και με τον συνάδελφο Πόλενσον και όλη του την ε, ομάδα, όλους τους συνεργάτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μοντραβέλ για όλα αυτά που μας είπατε και που απαντήσατε και στην ερώτησή μου. Ναι, πράγματι, αυτό είχα πει. Και επειδή όντω περνάει και ο χρόνος, να μην καθυστερήσω άλλο, να δώσω το λόγο στον κύριο Ροντρίγες από το Red Electrica. 10 λεπτά και εσείς παρακαλώ και παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να σας μιλήσω για την επαγγελματική μου ζωή. Θα προσπαθήσω με τη βοήθεια βέβαια και άλλων να συγχρονιστώ και να σας πω ότι εμείς έχουμε συνεργασία και με την Συρία και με τη Λιβύη και όλοι έχουν πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα, άλλο μέρος επαγγελματική μου η εμπειρίας είναι πώς θα συμπεριλάβουμε τις αλλακτικές πηγές ενέργειας σαν πηγή για ηλεκτρισμό. Αυτό γίνεται στη συνεργασία με το Μαρόκο. Μιλάμε συνέχεια για τον ε, ηλεκτρισμό. Ε, μιλάμε πολύ για δίκτυα. Μα το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελείται από αυτούς που παράγουν, από αυτούς που μεταφέρουν, φτάνουμε μέχρι και τους καταναλωτές. Όλα αυτά αποτελούν μέρος. Συζητώ συγγνώμη γιατί θα σας βάλω λίγο στη σημερινή πραγματικότητα. Στο, στη διαφάνεια αυτή βλέπετε το στόχο γύρω από τη Μεσόγειο. Το περίφημο Med Ring. Που όμως δεν είναι κλειστό. Υπάρχει Τουρκία-Συρία. 19-18 Σεπτεμβρίου η Τουρκία συνδέθηκε με το επιρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο συντονισμού, είναι χωρισμένα, που είναι η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Συρία, ο Λίβανος. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από το 1998 η Αλγερία, την Ισία και το Μαρόκο ε, βρίσκονται σε συντονισμό με μας. Πιο συγκεκριμένα η Λιβύη τώρα είναι αποκομμένη. Εξού η μαύρη γραμμή στην οποία αναφέρθηκε Άλμπερτ. Εδώ βλέπετε ανταλλαγές ενέργειας. Δεν είναι εύκολο να έχει κανείς πραγματικά νούμερα. Έχω χρησιμοποιήσει διάφορες πηγές, τις αναφέρω ποιες είναι αυτές. Αλλά για να έχετε μια ιδέα για το μέγεθος του συστήματος και για τις ανταλλαγές ενέργειας που γίνονται σήμερα μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Όπως βλέπετε, τα νούμερα δεν είναι πολύ μεγάλα. Πέρα από την περίπτωση του Μαρόκου. Το Μαρόκο εισάγει από την Ισπανία πολλή ενέργεια. Από πλευράς χωρών μας ΡΕΚ, τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά, αστεία. Για ποιο λόγο έχουμε τόσο χαμηλά ποσά, ποσότητες δηλαδή, δίκτυα αδύναμα δίκτυα. Και για να αποφύγουμε προβλήματα είμαστε σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Εδώ θα σας παρουσιάσω μία περίπτωση μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Γιβραλτάρ που πάει προς την βόρεια πλευρά των Πυρηναίων, βόρειος των Πυρηναίων. Υπάρχουν εδώ διάφοροι παράγοντες. Τεχνική, από τη μία, που είναι η δυνατότητα ανταλλαγών σε διεθνές επίπεδο, αλλά και περιορισμοί εσωτερικοί, εσωτερική ίδια τα συστήματα. Και το αριθμιστικό πλαίσιο, εντάξει, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και γι' αυτό πολύ, αλλά εγώ δεν θα επιμείνω για το αριθμιστικό πλαίσιο. Εδώ τι βλέπετε, βλέπετε ποια είναι η εξέλιξη της μεταφοράς αυτής. Βλέπετε τις χρονιές κάτω και πώς αυτή η δυνατότητα μεταφοράς μέσω των στενών του Γιβραλτάρ προς τα Πυρηναία προχωράει και αυξάνεται αλλά βέβαια μειώνεται εφόσον συμπεριληφθούν οι εναλλακτικές ενέργειες στην Ισπανία. Στην Ιβηρική Χερσόνησο. Τώρα θα κάνω διάφορες ε, υποθέσεις. Έτσι κι αλλιώς η φυσική είναι αυτή που είναι. Δεν αλλάζουν οι νόμοι της. Ας πούμε ότι έχουμε τρεις χώρες μέλη που έχουν ανταλλαγές μεταξύ τους. Μία από αυτές αρχίζει και λειτουργεί τα δικά της προγράμματα δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τι έχουμε, συμφόρηση. Πώς μπορεί να λυθεί αυτή η συμφόρηση? με περισσότερα δίκτυα, δίχως άλλο. Προσθέτουμε δίκτυα. Αυξάνονται τα δίκτυα. Όπως είπαμε, οι εναλλακτικέ πηγές ενέργειας ε, καταναλώνουν, απορροφάνε πολύ τα δίκτυα. Έπειτα, μέσω του ελέγχου της ε, παραγωγής. Ναι, αλλά πού γίνεται αυτός ο έλεγχος. Και πού, στο σύστημα Β, το Μαρόκο θα μειώσει την παραγωγή ολικής ενέργειας για να επιτρέψει μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας από την Τινησία, για παράδειγμα. Στην αρχική παρουσίαση θέλω να... Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, αλλά στο αφήσουμε για άλλη φορά. Έρχομαι στην επόμενη διαφάνεια. Όπως σας είπα, Βάζω ερωτήματα, αλλά προσπαθώ να δώσω και απαντήσεις. Ναι, διάφορες λύσεις που εμείς χρησιμοποίησαμε στην Ισπανία. η σωστή λειτουργία, χωρίς μείωση δηλαδή ούτε της ασφάλειας ούτε της ποιότητας, ε, των επιπέδων ασφάλειας και ποιότητας, απαιτούν κάποια πράγματα για τις εγκαταστάσεις όπου και αν βρίσκονται αυτές. Εκεί χρειάζεται βελτίωση και έχει γίνει βελτίωση βέβαια και για την ολική και για την ηλιακή. Έλεγχος. Ο έλεγχος ήταν στοιχείο κλειδί προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για τα 20 γιγαβάτ που έχουμε πει και για τα φωτοβολταϊκά και τη δικιά τους δυνατότητα έτσι όπως έχει αυτή στην Ιβηρική Χερσόνησο. Αλλά και από τη βιομηχανία χρειάζεται η σωστή απάντηση. Αν πάμε ακόμα παραπέρα, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των καταναλωτών. Πιο ευφύη αντιμετώπιση. Το βασικό βέβαια είναι οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς. Πρέπει εδώ να σας πω ότι από τότε που υπάρχουν ε, οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά τις εξελίξεις και έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το αποτέλεσμα δεν είναι πόσες γραμμές, πόσα χιλιόμετρα, πόσα καλώδια, πόσους αγωγούς χρειαζόμαστε, αλλά να ξέρουμε ποιος είναι ο χάρτης πορείας μας. Πού πάμε σε αυτούς τους ηλεκτρικούς αυτοκιν... ε, αυτοκινητοδρόμους κατά κάποιο τρόπο, διαδρόμους που θέλουμε να έχουμε για το 2050. Συμπεράσματα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα σημερινά δίκτυα δεν φτάνουν για την μαζική μεταφορά ενέργειας. Ούτε μεταξύ των δικών μας ευρωπαϊκών ε, συστημάτων, ούτε από τις χώρες ε, μέντα. Οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας από την άλλη μεριά χρειάζονται πολλά δίκτυα. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να γίνει χωρίς να μειωθεί το επίπεδο ασφάλειας των δικτύων μας. Πρέπει να καλυφθούν οι απαιτήσει. Παντού όπου έχουμε καταστάσεις. Πρέπει να υπάρχει επίσης έλεγχος και των ανώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των διαχειριστών δικτύων μεταφοράς. Πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα όσον αφορά την συμβατική παραγωγή και τέλος να υπάρχει αμοιβαιότητα, διαφάνεια και φυσικά να υπάρχουν μηχανισμοί πιστοποίησης για την δημιουργία ενέργειας από ανανόσιμες πηγές. Φυσικά πρέπει να το προστατεύσουμε το παιδί μας. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε, που μας ε, φώτισαν λιγάκι για το που βρίσκονται τα προβλήματα. Καλά. Μπορεί να περνάει ο χρόνος, αλλά θα δώσω την ευκαιρία στους συναδέρφους να υποβάλουν ερωτήσεις στους εισηγητές. Ο κύριος Τούρμες είναι ο πρώτος που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα θέσω μια ερώτηση. Μιλήσατε για χρήση όλων των πόρων. Για την πυρνική ενέργεια μετά τη Φουκουσίμα, ακόμα και αν η Γαλλία, η Αρεβά, η Ντεέφτα, ονειρεύονταν όλα αυτά, δεν νομίζω πια. Όμως, ε, ε, έχουν ηρεμήσει λίγο. Αυτό που με φοβίζει εμένα είναι ο άνθρακας. Θα ήταν καταστροφή αν το MedGrid χρησιμοποιηθεί τελικά ώστε να δοθεί η τεχνική δυνατότητα ένταξης πολύ μεγάλων μηχαλωμάτων ε, άνθρακα στην την ή στην Αλβανία γιατί τα εθνικά δίκτυα των χωρών είναι πολύ αδύναμα για αυτές τις πολύ βρώμικες μηχανές και άρα το γεγονός ότι εμείς φτιάχνουμε καλώδια θα καθιστούσε τεχνικά δυνατή αυτή την ε, οικολογική καταστροφή. Θα πρέπει λοιπόν να τοποθετηθείτε για το ποια είναι η προτεραιότητά σας σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί να καταστούν δυνατές οι εισαγωγές άνθρακα προς την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι κάτι που εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ήδη έχουμε ξεκάθαρη θέση γι' αυτό και νομίζω πως το γνωρίζετε κι εσείς, ότι στα έγγραφα για τις υποδομές, στην ανακοίνωση, υπάρχουν δύο παράγραφοι που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν αυτό θα το φροντίσουν. Και για τη μελλοντική μας συνεργασία λοιπόν θα ήταν καλό αν μπορούσατε κάπως να με καθησυχάσετε για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ άλλους αν σε το λόγο και μετά εσείς. Ευχαριστώ Τερέζα. Ε, και εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Αντράν. Ο Ισπανός συνάδελφος μίλησε για το πακέτο κλίμα-ενέργεια και εισήχθη ένας μηχανισμός για την ε, καθαρή ανάπτυξη, ένας μηχανισμός ε, ε, καθαρής ανάπτυξης που επιτρέπει στα μέλη να χρησιμοποιούν το 3% των εκπομπών τους αν βοηθήσουν τρίτες χώρες, ώστε αυτές να αναπτύξουν παραγωγικές μονάδες πιο αποτελεσματικές από την άποψη της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων στην ανανεώσιμη ενέργεια. Ήθελα λοιπόν να σας θέσω το ερώτημα. Υπάρχει τέτοιο είδους επένδυση σε εσά. Ξέρω πως ψάχνετε επενδυτές. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια πιθανή πηγή χρηματοδότησης. Δεύτερη ερώτηση. Έπειτα, για αυτό το πακέτο για το κλίμα. Έχουμε χώρες όπως το Λουξεμβούργο, πουχού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν χώρες που έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το ποσοστό το 3% και αν, γιατί δεν αν όχι γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ, αν κατάλαβα καλά, είπε πως ο μηχανισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται αρκετά. Αυτή η δυνατότητα το 3% υπάρχει. Γιατί δεν χρησιμοποιείται και εφόσον υπάρχει ρήπανση, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 3% ρήπανσης για να το αντισταθμίσουμε. Γιατί δεν το χρησιμοποιούμε. Ευχαριστούμε για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη προς τον κύριο Μαντραβέλ, ο οποίος θα πάρει και πρώτο το λόγο, μετά ο κύριο Σαντουράνη και τέλος ο κύριος Ροντρίγες. Σας ακούμε. Κύριε Μαντραβέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ θα απαντήσω μόνο στο ερώτημα του κύριου Τούρμες, γιατί εκεί σε αυτό είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Και άλλωστε η ερώτηση αφορούσε άμεσα το MedGrid. MedGrid. Το MedGrid φυσικά και δεν θα ευνοήσει τη δημιουργία ε, εργοστασίων που ρηπαίνουν. Αλλά όταν φτιάχνουμε ένα δίκτυο μεταφοράς, τα διάφορα κομμάτια του παίρνουν τον ηλεκτρισμό που προέρχεται από ένα εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας ή ε, εργοστάσιο που χρησιμοποιεί άνθρακα και από τη στιγμή που φτιαχτεί αυτό το δίκτυο μπορεί να μεταφέρει κάθε είδους ηλεκτρισμό ακόμα και πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια. Ξέρω ότι δεν χρειάζεται να το λέω αυτή τη στιγμή γιατί δεν είναι πολιτικό ορθή η πυρηνική ενέργεια αυτή την περίοδο αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αλήθεια. Τώρα εξαρτάται αν η Κομισιόν ή το Ευρωκοινοβούλιο θα επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο, θα εξαναγκάζουν τις χώρες να συνδεθούν μεταξύ τους Ισπανία-Γαλλία, Γαλλία-Γερμανία. Αυτά όλα δεν έχουν σχέση με το είδος της, της ηλεκτρικής ενέργειας που θα μεταφέρεται μέσα από αυτές τις νέες συνδέσεις. Άρα λοιπόν αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το MedGrid φυσικά και δεν πρόκειται να ευνοήσει τέτοιου είδους ε, εγκαταστάσεις ε, ηλεκτροπαραγωγικές που ρηπαίνουν, αλλά το δίκτυο, το δίκτυο εμείς θα φτιάξουμε. Το δίκτυο θα μεταφέρει ηλεκτρική, ηλεκτρισμό από όπου και αν προέρχεται για να ευνοήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι αλλά και να, ε, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια ε, ανεφοδιασμού και τις συναλλαγές σε ηλεκτρισμό προς όλες τις κατευθύνσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Ντράνη, δεν ξέρω τι έχετε να απαντήσετε. Θα αφήσει το Μαρόκο να περάσει ενέργεια εναλλακτική που έχει παραχθεί στην την Ισία, για παράδειγμα. Τι λέτε. Δύσκολο να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, νομίζω ότι ασχολούνται με την ηλεκτρική ενέργεια είναι πιο προχωρημένοι. Ε, γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα μερικές φορές από τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί έχουν λόγο όταν πρόκειται για τη διατήρηση, τη βελτίωση ενός δικτύου, δεν υπάρχει θέμα εκεί αλλά για την κινητοποίηση πόρων στο Βαρσαζάτ να ξέρετε ότι έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι πόροι στήριξης που υπάρχουν σήμερα από δωρές, αλλά και από άλλες συμβατικές μορφές χρηματοδότησης, έτσι όπως προβλέπονται από τους δωρητές σε διεθνές επίπεδο. Ο μηχανισμός ε, η καθαρή ανάπτυξη επίσης συνεισφέρει. Το 3% δεν μου λέει τίποτα έτσι από Θα προσπαθήσω να κοιτάξω μήπως υπάρχει κάτι άλλο για να μην σας λέω ανοησίε. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ροντρίγες τώρα. Σας ικανοποιεί η απάντηση του κύριου Μπράνε ε, βάλαμε, σαν παράδειγμα, βάλαμε σαν παράδειγμα το Μαρόκο και την Τινησία. Γιατί για να βγούμε λιγάκι από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα ήταν πιο εύκολο εγώ να σας πω εγώ στην Ισπανία πρέπει να μειώσω την νεολική μου ενέργεια για να επιτρέψω όλες τις μορφές ενέργειας να περάσουν. Ήθελα να αποφύγω το ευρωπαϊκό πλαίσιο και γι' αυτό έβαλα το παράδειγμα το άλλο. Αλλά να προσθέσω ότι στόχοι καταπολέμησης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα περνάνε μέσα από την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή αποτελεί το μέσο για να πετύχουμε το στόχο μας. Τώρα και εγώ ως διαχειριστής δικτύου μεταφοράς, ως οδηγός εντό αγωγικών του λεωφορείου αυτού που ονομάζεται ηλεκτρικό σύστημα, τι κάνω προσπαθώ να το οδηγήσω με τον πιο ασφαλή τρόπο και με επίπεδα ποιότητας, έτσι όπως απαιτεί μια κοινωνία που εξαρτάται από τον ηλεκτρισμό και ανεξάρτητα από το αν οι ρόδες που έχω είναι η μία από ξύλο, η άλλη από πλαστικό, η άλλη από δεν ξέρω εγώ τι. Πρόεδρος, καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, εδώ τελείωσε το δικό μου έργο. Ευχαριστώ πολύ όλους τους εισηγητές για τις παρουσιάσεις τους. Και ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας εδώ. Και τώρα παραχωρώ την Προεδρία στον συνάδελφο Τούρμες. Uh, so, uh, I, propose that we, immediately. Uh, Προτείνω να ξεκινήσουμε αμέσως. One problem is that at six o'clock I will have to to leave because I, have. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σύντομα. Σε κάποια φάση θα πρέπει να λείψω. Γιατί πρέπει να συμμετέχω σε κάτι διαπραγματεύσεις για το REMIT, για τη διαφάνεια στην αγορά ηλεκτρισμού, που είναι επίσης σημαντικό θέμα. Δεν ξέρω, πιθανότατα κάποιο από τη γραμματεία θα προεδρεύσει στην υπόλοιπη συνεδρίαση. Κανονικά θα έχετε 10 λεπτά ο κάθε ομιλητής. Αν μπορείτε να τα πείτε λίγο πιο γρήγορα, θα ήταν ευκταίο. Παρακαλώ, η κυρία Μαρκέσης είναι μόνιμη εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ενεργειακής Πολιτικής και ασχολείται και με το ΙΜΕΝΤΑ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την εισήγηση. Θα ήθελα να τονίσω πόσο ενδιαφέρουσα είναι αυτή, ε, ε, αυτή εδώ η εκδήλωση. εντάσσεται στο, εταιρική, στο πλαίσιο της εταιρική σχέσης για την Μεσόγειο για τη διαχείριση της ανανεώσιμη, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά συνδέονται με το σενάριο 2050 για την Ένωση με νέες εταιρικές σχέσεις με την προϋπόθεση ότι θα έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες προπτικές για την εισαγωγή ηλεκτρισμού. Επίσης αυτό έρχεται μετά από την ανακοίνωση για το μέλλον της ε, πολιτικής γεννήσης που υιοθετήθηκε πιο πρόσφατα και που πάλι τονίζει την ανάγκη για ορισμό νέων ε, προγραμμάτων συνεργασία και ανάπτυξη με του νότιου γειτονέ μα και έπειτα προηγείται μια επερχόμενη ανακοίνωση, όπου περιγράφεται η στρατηγική για την εξωτερική διάσταση της ενεργειακή πολιτικής της ΕΕ όπου μεταξύ άλλων επίσης ε, θα δούμε τις δυνατότητες για ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων ε, όσον αφορά τη σταδιακή συμμετοχή στην ενεργειακή αγορά της ε, Ένωσης. Οποτεδήποτε γίνεται λόγο για ενέργεια στην Νότιο Μεσόγειο ή για την ανανεώσιμη ενέργεια κυρίω θα πρέπει να έχουμε μονίμω υπόψη μα κάποια στοιχεία. Καταρχήν, οι γείτονέ μα ε, περνούν άνευ προηγουμένων αλλαγέ, σαν δημογραφική ανάπτυξη, κοινωνικέ μεταρρυθμίσει ε, και παντού οι πληθυσμοί ισχυρίζονται το δικαίωμά του στη συμμετοχή στην οικονομική και πολιτική ζωή τη χώρα του. Επίση, ε, υπάρχει μεγάλη αύξηση πληθυσμού στις χώρες αυτές. Ταυτόχρονα καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια κατά κεφαλήν από ό,τι εμείς. Ίσως και τρεις φορές λιγότερο από ό,τι εμείς, σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Αλγερία για παράδειγμα. Και οι οικονομίες τους αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι οικονομίες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Για όλα αυτά σε όλους αυτούς τους λόγους η κατανάλωση ενέργειας θα διπλασιαστεί εντός λίγων ετών. Ακούσαμε τον προηγούμενο μιλητή ότι θα πολλαπλασιαστεί επί τέσσερα μέχρι το 2030. Τεράστια πρόκληση αυτή, αλλά για εκείνους αλλά και για μας, διότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι οι επιλογές οι επενδυτικές που θα γίνουν εκεί σαφώς θα επηρεάσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πολιτική προώθηση αναθεώσιμων πηγών ενέργειας στις χώρες της Νοτίας Μεσογείου θα πρέπει να ξεκινήσουν μέσω της κάλυψης των άμεσων αναγκών της περιοχής. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, γιατί υπάρχουν διάφορα πλαίσια που υπάρχουν. Όπως ξέρετε υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και τις νότιες χώρες Μεσογείου και καλύπτεται από πολιτικής άποψη από ισχύουσε ισχύουσες ε, συμφωνίες σύνδεσης καθώς και για το ειδικό, από το ειδικό μνημόνιο συνεννόηση για την ενέργεια. Για την ώρα στηρίζουμε κάποιες ε, πρωτοβουλίε περιφερειακή συνεργασία, όπως η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς στο Μαγκρέμπ καθώς ε, και στο Ισραήλ Επίσης, ε, δίνουμε σημαντική στήριξη στους προπολογισμού για τομεακές μεταρρυθμίσεις σε πολλές από τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, καθώς και διεξάγουμε διάφορα προγράμματα τοπικής ε, συνεργασίας για την ανανεώσιμη ενέργεια και την επάρκεια ενέργειας. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα σας δώσουν τις λεπτομέρειες για τα σημαντικά δάνεια και προγράμματα που έχουν διατεθεί υπό το ΦΕΜΙΠ. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία που προσδίδουμε στην στήριξη που δίνεται από το μέσο το επενδυτικό μέσο στην ε, γυρνίαση. Τώρα όσον αφορά την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, συχνά λέγεται ότι οι εξαγωγές ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα επέτρεπε τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στις χώρες της Νότιας Μεσογείου. Ωστόσο, εάν λάβουμε τον αν δούμε τον ορίζοντα 2020, δεν μπορούμε να δούμε ένα σαφές επιχειρηματικό ρυθμό για την ώρα. Επί τη βάση των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, η Ένωση φαίνεται να ξεπερνά κάπως τον στόχο του 20% για το 2020 και με τη βάση των πληροφοριών που δίνουν τα κράτη-μέλη για το εθνικό τους πλάνο δεν αναφέρουν σημαντικές εισαγωγές από τις χώρες της Νοτιάς Μεσογείου. Μάλιστα, η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στις νότιες χώρες δεν έχει πρόσβαση στα καθεστώτα επιδότησης που δημιουργούν τα κράτη-μέλη και χωρίς τέτοιες επιδοτήσεις η ηλιακή ενέργεια ακόμα και αν λάβει κανείς υπόψη την υψηλότερο, τον παράγοντα υψηλότερης ακτινοβολίας δεν θα ήταν συμβατή για την, ε, ενέργεια, για την αγορά ενέργειας στην Ένωση στα επόμενα χρόνια. Μιλάω για μέχρι το 2020. Άρα λοιπόν οι εισαγωγές ηλεκτρισμού μπορεί να είναι συμβατές μετά από το 2025 ανάλογα με διάφορους παράγοντες, την εξέλιξη της τεχνολογίας δηλαδή, την τιμή του άνθρακα και την τιμή της ορυκτής ενέργειας, των ορυκτών καυσίμων και αυτό όμως είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς είναι πιο δύσκολο να χρηματοδοτηθούν οι ανανεώσιμες, ιδιαίτερα για την ηλιακή ενέργεια στις νότιες χώρες της Μεσογείου, λόγω του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου. Υπάρχει μεγάλη αύξηση της ζήτησης, επενδυτική κίνδυνη, κοινωνική αστάθεια, για να αναφέρω μόνο κάποια ως παράγοντες. Ορισμένες χώρες όμως θα μπορούσαν να, να, να δρομολογήσουν τις επιδοτήσεις που παίρνουν οι ορυκτές, ε, τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες ε, ενέργειες. Βέβαια αυτό θα σήμαινε θαραλές αποφάσεις για αύξηση των τιμών του ηλεκτρισμού, πράγμα το οποίο δεν είναι διόλου προφανές σε αυτή τη φάση. Εν τω μεταξύ αρκετές νότιες χώρες έχουν αποφασίσει να αναπτύξουν τις ανανεώσιμες ενέργειες μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών τους προγραμμάτων ανάπτυξης. Τα εργαλεία μας θα πρέπει να επαναξιολογηθούν γιατί ούτε η τεχνική βοήθεια ούτε το άρθρο 9 δεν θα αρκέσουν για να γίνουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Γι' αυτό η πρόταση της Κομισιόν για εκκίνηση συζήτησης για το πιθανό περιεχόμενο μιας ε, συνεργασίας Ένωσης Μεσογείου για τη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα σήμαινε επενδύσεις στο Νότο, θα σήμαινε μελέτη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Μια τέτοια συνεργασία θα πρέπει να καθοριστεί μέσω ενός προγράμματος με τους εταίρους μας. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε με τα κράτη-μέλη καθώς και με τη διεθνή χρηματοδοτική κοινότητα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Οι συζητήσεις συνεχίζονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο και διάφορους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό σχετίζεται και με το θέμα που αρχικά θύχθηκε στο πρώτο πάνελ και που σχετίζεται με το upstreaming της ενέργειας και τη ανάπτυξη των διαφόρων πηγών ενέργειας. Ε, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, πολύ ε, που ήσασταν και σύντομοι. Ε, έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ τον κύριο Walters κοντά μας. Ε, γνωριστήκαμε στη διάσκεψη της Σεβίλης. Ε, η Παγκόσμια Τράπεζα παίζει πολύ ε, ενεργό ρόλο. Μήπως μπορείτε παρακαλώ να μας κάνετε μια ενημέρωση σχετικά με το πού βρίσκεστε, τι επιτυχία είχατε σχετικά με την χρηματοδότηση μεγέθους ενός δισεκατομμυρίου, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ σήμερα και για την ωραία εισαγωγή σας. Θα πρέπει να ανταγωνιστώ την πόλα όσον αφορά την συντομία. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι σύντομος διότι πολλά υπόθηκαν ήδη. Ε, θα... Ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο από το Μαρόκο για την ομιλία του, διότι ε, συμφωνώ μαζί του τουλάχιστον κατά 100%. Συχνά λέω στον κόσμο ότι η η ηγεσία του Μεσογειακού Σχεδίου Λιακής Ενέργειας έχει περάσει στο Μαρόκο, στο Ραμπάτ και ότι αυτό αποτελεί στρατηγική πρόκληση για την ε, Ευρώπη ε, αλλά και για την ε, Βόρεια Αφρική. Είναι μια πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ε, αναφερθώ στην, ε, συγκεντρωμένη στην πρωτοβουλία για την συσσωρευμένη ηλιακή ενέργεια. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι εταίρος ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων, την Ισλαμική Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και, άλλες, καθώς και άλλους διμερείς φορείς ανάπτυξης από την Ευρώπη και αλλού. Πρωτού όμως φτάσω σε αυτό, θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις σχετικά με τη συσσωρευμένη ηλιακή ενέργεια. Η πρώτη είναι ότι ο κόσμος ε, σαφώς αναζητά περισσότερες λύσεις ε, για ενεργειακές πηγές ε, 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ορικτές ε, χωρίς ορυκτά καύσιμα. Αυτό θα είναι σημαντικό ε, όσον αφορά την προστασία του κλίματος και την ε, ασφάλεια εφοδιασμού. Έχουμε την πυρηνική ενέργεια, τη γεωθερμική ενέργεια. Σίγουρα πρέπει ο κατάλογος να είναι μακρύτερος, θα πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος και για να γίνει αυτό θα πρέπει να είμαστε προορατικοί φιλόδοξη και να ε, στηρίξουμε τις διάφορες τεχνολογίες. Σε μία λύση ε, πολλά υποσχόμενη στο μενού είναι η συσσωρευμένη ηλιακή ενέργεια, όχι μόνο λόγω της ε, διαθεσιμότητας της δωρεάν ηλικής ενέργειας στις ρήμους, αλλά και επειδή η αποθήκευση της θερμότητας ε, φαίνεται να είναι πιο ενδιαφέρουσα, πιο οικονομική από την ε, αποθήκευση ε, ηλεκτρισμού. Είναι λοιπόν μια τεχνολογία που υπόσχεται πολλά. Η ηλιακή ενέργεια είναι μεταβάσιμη ενέργεια. Πολύ μικρό κομμάτι έχει διανοητικά δικαιώματα, λιγότερο από το 10% της αξίας. Οι περισσότερες χώρες που έχουν ε, ε, οικοδομικό, οικοδομικό τομέα, ε, γυαλιού ή ατσαλιού μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να υιοθετήσουν τις τεχνολογίες αυτές. Είναι πολύ δύσκολο να υπερτιμήσουμε την σημασία της ε, της τεχνολογίας αυτής. Ε, ήταν σημαντική στο παρελθόν, ε, πόσο μάλλον τώρα ε, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Θα ήθελα να αναφερθώ στη σημασία της ορμένης ηλιακής ενέργειας για πέντε χώρες στο, στην περιοχή. Μία ε, αρκετά με τριοπαθής ε, μελέτη αναφέρεται σε ε, δημιουργία πολλών ε, θέσεων εργασίας στις χώρες αυτές. Όλα βέβαια εξαρτώνται από τον όγκο των Μεγαβάτε που θα ε, δημιουργηθεί. Ε, άλλη παρατήρηση για τη συσσωρευμένη ηλιακή ενέργεια είναι ότι είναι μια τεχνολογία που παρότι σε μεγάλο βαθμό έχει αποδείξει την αξία της από πλευράς τεχνολογίας υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας ε, τις οποίες δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα. Ε, όπως είπε ο κύριος Ευανζόνη, είναι το προβληματικό μας παιδί που δεν έχει μάθει ακόμα να περπατάει. Το κόστος είναι υψηλό επειδή η ζήτηση είναι μικρή ε, και η ζήτηση είναι μικρή επειδή το κόστος ε, είναι ψηλό. Για να ξεπεράσουμε λοιπόν το όριο θα πρέπει να υπάρξουν ε, σημαντικές επιδοτήσεις μέχρι να γίνει ανταγωνιστική τεχνολογία αυτή. Μαζί με τους άλλους φορείς ανάπτυξης λοιπόν που σας ανέφερα έχουμε δημιουργήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης για χίλια ΜΒ συσσωρευμένης ηλιακής ενέργειας ε, στην ε, Μεσόγειο, καθώς ε, και δίκτυα διαβίβασης ώστε να βοηθήσουμε την εξαγωγή. Το κόστος είναι, γενικά, είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Χίλια ΜΒ από μόνα τους δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι είναι εφικτό αυτό, ότι γίνεται κάτι συγκεκριμένο και είναι, ελπίζουμε, κάτι το οποίο θα οδηγήσει ε, σε, ε, σε περαιτέρω τέτοια προγράμματα για να μειωθεί περαιτέρω το κόστος. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, ε, τόσο γρήγορα που έχουμε εντυπωσιαστεί όλοι μας. Έχει βρει χρηματοδοτική υποστήριξη, όπως κάποιος ανέφερε όμως πριν, μπορεί να χρηματοδοτηθούν όλα τα προγράμματα αυτά. Το σημαντικό όμως είναι η όροι της χρηματοδότησης ε, και αυτό οδηγεί σε δύο σημαντικά ε, θέματα. Πρώτον, από πού θα δοθεί χρηματοδότηση και ε, ε, σίγουρα η χρηματοδότηση για την προστασία του κλίματος από το, το πρωτόκολλο του Κιώτο μαζί με τις ε, συμφωνίες ε, Κανκούν, τέτοιου είδους χρηματοδότηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές. Ξεκινάμε με τα 6 δισεκατομμύρια τα οποία ανέφερα. Έχουμε μια επιδότηση από το Ταμείο Καθαρών Τεχνολογιών ε, περιμένουμε όμως και άλλα. Και η άλλη πηγή χρηματοδότησης ε, είναι αυτά τα οποία ήδη συζητήσαμε ε, σήμερα. Οι εξαγωγές δηλαδή προς την Ευρώπη και σε αγορές πράσινης ενέργειας. Ε, τα, ακούσαμε όλα τα σχετικά, το άρθρο 9 και το ε, Μεσογειακό Σχέδιο Ελληνικής Ενέργειας. θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν πιο συγκεκριμένα. οι πρώτες εξαγωγές ήδη πραγματοποιούνται είδαμε πολλές ε, παρουσιάσεις σε πολλές διασκέψεις. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις μονάδες παραγωγής ε, ώστε ο κόσμος να πιστέψει ε, ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό. Μπορεί να μην φτάσουμε το 20% το 2020, το 20% είναι ο στόχος το 2020 πλησιάζει, είναι πολύ κοντά, θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο μακροπρόθεσμα, να δούμε τις ε, μειώσεις εκπομπών ε, τις, ε, με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει με την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων, ειδικά η υποστήριξη που θα βοηθήσει στο ξεκίνημα, δηλαδή με συμβάσεις εξαγωγών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Τζόναθαν. Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα το απόγευμα ήταν η αξιολόγηση του κινδύνου, διότι ε, ο κόσμος ε, κινείται από την οικονομία. Ε, έχουμε μέσα για να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτόν και τους τόχους στα δάνεια. Βρισκόμαστε σε εξαιρετική θέση, διότι έχουμε δύο εκπροσώπους εδώ του, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, μπορείτε λοιπόν να μοιραστείτε το ε, δεκάλεπτο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Αυτό που θέλω είναι ουσιαστικά να χτίσω πάνω σε αυτά που συζητήθηκαν σήμερα και πάνω στις παρουσιάσεις των άλλων για να καταλήξω σε τέσσερις παρατηρήσεις από την δικιά μου την πλευρά και να σας δώσω μια ιδέα για το τι κάνουμε στο Μεσογειακό Solar Plan. Πρώτον, πέρυσι είχαμε μια χρονιά κρίσης με 2,6 δις επένδυση στις χώρες εταίρους της Μεσογείου. Τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε χρηματοδοτήσει με 12 δις ευρώ το οποίο κινητοποίησαν άλλα 30 με 35 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Κάτι το οποίο κάνει το IB τον ε, μεγαλύτερο εταίρο. Κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ξέρει και η Ευρώπη πρέπει να ξέρει και να είναι περήφανη γιατί ουσιαστικά είναι η τράπεζα εκείνη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δηλαδή, η οποία έχει κάνει τόσα πολλά. Εξαρτώμεθα κατά πολύ από εσά. Διότι εμείς δεν κάνουμε πολιτική, παίρνουμε πολιτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Οπότε ακολουθούμε τις δικές σας εντολές, εξαρτώμεθα από εσά. Ξέρετε μάλιστα ότι εσείς διαπραγματεύεστε το μέλλον των δικών μας εντολών. Είμαστε δηλαδή στα δικά σας χέρια, εσείς μας λέτε τι να κάνουμε, τι να κάνουμε περισσότερο, τι να αλλάξουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακολουθούμε τις δικές σας προτεραιότητες λοιπόν, αυτές που εσείς μας έχετε μεταφέρει και η προτεραιότητά σας είναι ενέργεια, ανανόσιμες πηγές ενέργειας στις μεσογειακές χώρες. Από τα 12 λοιπόν δις ε, στα οποία αναφέρθηκα, το 1,5 δις πήγε στην ενέργεια και για τις ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας έχουμε ως στόχο το 50%. Απόλυτα φυσιολογικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο μεγαλύτερος ε, ε δωρητής με 6,2 δις πέρυσι συνολικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ότι κάναμε, το κάναμε και με προγράμματα που αξίζει να το αναφέρουμε. Αναφέρθηκε κάπου η κινέζικη τεχνολογία. Ε, λοιπόν, είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη στην τεχνολογία έρευνας και καινοτομία, ώστε να έχουμε έναν άσωστο στο μανίκι μας. Δεν είναι καινούργια αυτά τα θέματα για την ΕΤΕ. Είχαμε προγράμματα ηλιακή ενέργεια στην Ισπανία. Είναι κάτι το οποίο πέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να ξέρετε, το οποίο προώθησε με την νομοθεσία την κατάσταση έτσι ώστε να επενδύσουν οι χώρες στην ηλιακή ενέργεια. Άρα έχουμε ήδη κάποια εμπειρία και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης. Το τέταρτο σημείο μου έχει να κάνει με το μέλλον και την αναπτυξιακή βοήθεια. Εδώ πρέπει να σας πω, μια που έχω δουλέψει και στην Παγκόσμια Τράπεζα, που είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο που έχει ασχοληθεί και με τη Λατινική Αμερική και με την υποσαχάρια Αφρική, να σας πω ότι οι χώρες της Βόρειας Αφρικής δεν χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Αν μιλήσετε για, με, το, με το Λίβανο, το Μαρόκο κτλ. δεν θέλουν φιλανθρωπία. Αυτό που θέλουν είναι να τους παίρνουμε σοβαρά σαν εταίρους επενδυτές. Θέλουν επενδυτικές ευκαιρίες. Και οι χώρες αυτές που ποτέ δεν θα είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει αυτό ακριβώς που κάναμε εμείς τα τελευταία 50 χρόνια μας μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι περιφερειακές ευρωπαϊκές χώρες να έρθουν στο ίδιο οικονομικό επίπεδο με την υπόλοιπη Ευρώπη, με τη Δυτική Ευρώπη. Αυτές οι ευκαιρίες θέλουν. Αυτό θέλουν λοιπόν αυτές οι χώρες και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το μέσον ακριβώ που διαθέτει η Ευρώπη για να το κάνει αυτό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το άρθρο 9, στο οποίο αναφέρθηκε και η Γραμματεία τη Ένωση ε, για την Μεσόγειο, βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε συζητήσει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη Γραμματεία τη Ένωση για τη Μεσόγειο μετά από δικέ σα εντολές για να καταλήξουμε σε οικονομικέ λύσει προκειμένου να επιταχύνουμε τι επενδύσει. Αυτά. Ευχαριστούμε Γιάννη και Πρόεδρε. Όπως είπε και ο συνάδελφος, η ενέργεια είναι προτερότητα για την ΕΤΕ. Πάνω από 1,4 ε, δις επενδύσαμε στην Μεσόγειο. Η προτερότητα αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο με το πρόγραμμα για ηλιακή ενέργεια την Μεσόγειο. Το 2008 το Συμβούλιο Κοφίν έδωσε εντολή στην ΕΤΕ να συντονίσει ε, την ε, οικονομική εφαρμογή του Mediterranean Solar Plan. Ήταν λοιπόν προτερότητά μας. Συνεργαστήκαμε με την Ένωση για την Μεσόγειο και καταλήξαμε στο πρόγραμμα δράσης μας. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο σας παρουσιάστηκε από μακρό. Αυτό όμως που έχω να σας πω είναι ότι ως ΕΤΕ την εντολή μας την πήραμε από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και την πήραμε πάρα πολύ σοβαρά με διάφορες δράσεις. Χρηματοδοτήσαμε καταρχήν μια μελέτη για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας στην περιοχή. Στόχος της μελέτης ήταν να εντοπίσει συγκεκριμένα προγράμματα σε όλες τις 9 χώρες εταίρους μας στη Μεσόγειο και καταλήξαμε σε 85 τέτοια προγράμματα. Αυτό ήταν ε, το πρώτο, η πρώτη μας ε, βάση για να προχωρήσουμε με το Mediterranean Solar Plan. Μετά από τη μελέτη αυτή που έγινε από το Trust Fund που διαχειρίζεται η ΕΤΕ, δουλέψαμε σε συνεργασία με εταίρους μας από τον οικονομικό κόσμο για να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτή την εποχή ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα του Μαρόκο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Τζον. Γιατί συγχρηματοδοτείται από την ΕΤΕ, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από αναπτυξιακές αφρικανικές τράπεζες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εμείς την θέση λειτουργία των προγραμμάτων αυτών. Συνεργασία με τους άλλους οικονομικούς παράγοντες. Πέρα από αυτό, όμως υπάρχουν και άλλα συγκεκριμένα προγράμματα στην περιοχή που εξετάζονται από την ΕΤΕ. Αιωλική τεχνολογία, ηλιακή τεχνολογία και μιλάμε για όλες τις χώρες. Έχουμε ήδη διάφορα προγράμματα υπόψη στην Ιορδανία, το Μαρόκο, την Αίγυπτο. Το καθήκον αυτό λοιπόν που αναλάβαμε από το Συμβούλιο Κοφίν το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Τέλος. Δεν είμαστε μόνοι μας. Συμφωνούμε και εμείς για το ότι χρειάζεται στήριξη, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο εφαρμογής, γιατί κάποιες τεχνολογίες είναι στην αρχή ακόμα. Άρα χρειαζόμαστε οικονομική στήριξη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι κάτι που αποφασίζεται κάθε οικονομικό έτος και με την Παγκόσμια Τράπεζα και με διμερείς συμφωνίες και με άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα συζητάμε. Έτσι πιστεύουμε ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι του SP. Προτού να προχωρήσουμε στον ε, δόκτωρα Φουκέ, στην ε, δόκτωρα Φουκέ, ε, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η, δική σας γνώμη, τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε εμείς τα πρώτα μεγάλα προγράμματα. Και ε, ε, συμφωνώ με το μήνυμά σας αυτό. Θα πρέπει φυσικά να γίνουμε πιο ορατοί. Υπάρχει το άρθρο 9, υπάρχουν άλλα θέματα. Ε, τι μέσο όμως μπορεί να παράσχει η Ευρώπη για να μειώσει ε, τους στόκους των δανείων. Υπάρχει κάτι που εμείς οι πολιτικοί πρέπει να καταλάβουμε. Να διασαφηνίσω ότι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους αυτή τη στιγμή στην περιοχή που εμποδίζει ε, τους επενδυτές είναι ο, πολιτικός κίνδυνος ε, μετά από όσα ε, συνέβησαν ε, στην, στις χώρες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όμως έχει εφαρμόσει το καταπληκτικό αυτό μέτρο που είναι η κάλυψη του πολιτικού κινδύνου. Και ε, το, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ στη Μεσόγειο το μέσο αυτό. Να σα εξηγήσω τι ακριβώ συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ε, που μα ρωτούν πότε θα αρχίσουμε να δουλεύουμε στη Λιβύη. Στη Λιβύη δεν χρειάζονται χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έχουν ένα σωρό χρήματα εκεί. Θα χρειαστούν όμως την κάλυψη πολιτικού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εάν ε, λοιπόν ε, το Κοινοβούλιο και ε, ομαλοποιηθεί η πολιτική κατάσταση και συμφωνήσει το Κοινοβούλιο για τις επενδύσεις στη Λιβύη, τότε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι ακραία η περίπτωση που σας λέω, αλλά τότε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παράσχει την κάλυψη του πολιτικού κινδύνου. Συνήθω Συνήθως οι χώρες δεν θέλουν να ε, αντιταθούν σε μια επένδυση που έχει την σημαία, τη σφραγίδα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ότι δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις τους με την Ευρώπη. Είναι λοιπόν ε, μια επένδυση με πολύ ε, ισχυρή δύναμη μόχλευσης. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω την, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατηρήσει την κάλυψη αυτή. Υπάρχουν βέβαια άλλοι κίνδυνοι, εμπορικοί, ε, νομικοί, ε, επενδυτικοί κλπ. Αυτή τη στιγμή η σχετική γραμματεία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει μια ομάδα εργασίας που εξετάζει τους διάφορους κινδύνους και μια εξαιρετική ιδέα είναι να ε, υπογράψει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και οι χώρες εταίροι μια συμφωνία πολιτική σχετικά με τους όρους που θα πρέπει να σεβαστούν οι χώρες αυτές για να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρήματα. Εάν λοιπόν η Κομισιόν και οι χώρες εταίροι υπογράψουν τέτοια σύμβαση, τότε σε όλες τις συμβάσεις θα γράφει ότι πρέπει οι χώρες εταίροι να σεβαστούν τη συμφωνία αυτή για να έχουν πρόσβαση στα χρήματά μας επειδή είμαστε ε, φορές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, περνάμε τότε στις λεπτομέρειες του άρθρου 9, τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους Ενό άρθρου 9 εάν δεν είναι καλά διατυπωμένο και έχουμε ε, τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας την κυρία Φουκέ που εργάζεται μήνες, μηνες από χρόνια πάνω στο θέμα αυτό. Μήπως μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μουράν, κυρίες και κύριοι, Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Υπάρχει ένα PowerPoint, αλλά δεν θα σας το παρουσιάσω. Θα σας μιλήσω για δύο-τρεις από τις διαφάνειες που έχω εδώ μπροστά μου. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να πω ως νομικός, θα σας πω ότι εργάζομαι με συναδέλφους σε αυτό το τομέα εδώ και πολύ καιρό. Η δουλειά είναι υπό εξέλιξη. Ακόμα μαθαίνουμε με τα διάφορα κράτη-μέλη με τα οποία συνεργαζόμαστε. Με ανθρώπους σαν τον Κλοντ και άλλους αλλά για να, θέλω να καταστήσω κάτι σαφές εξ αρχές, ότι είναι πολύ καλό να ε, μπορούμε να πούμε ότι ναι, πρέπει να κάνουμε ένα πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα για να αποδείξουμε ότι λειτουργεί, αλλά και να σπάσουμε κάποιους γόρδιους δεσμούς που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αφρικής, αλλά και τις σχέσεις εντός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να αναλύσουμε είναι να απο... καθυλώσουμε το άρθρο 9. Είναι εξαιρετικά πολιτικοποιημένο και υπερτιμημένο στο τι θέλει κανείς να κάνει με αυτό το άρθρο. Και όπως έχει ήδη το άρθρο 9 είναι κομμάτι τριών μηχανισμών ευελιξίας στην ε, οδηγία για την ανανεώσιμες ενέργειες. Στόχος της οδηγίας είναι να φτάσουμε μήνυμο 20% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός της Ένωσης μέχρι το 2020. Και Έγινε και η συζήτηση ότι προ χάρη αποτελεσματικότητα και απόδοση και κόστος ωφέλειας ορισμένα μέλη που το επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό ευελιξία. Πρέπει να το πούμε δηλαδή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την οδηγία θέλουμε να αλλάξουμε τα συστήματά μας και να χρησιμοποιήσουμε την ανανεώσιμη ενέργεια. Ένα εργαλείο είναι το εργαλείο της ευελιξίας και το άρθρο 9 είναι κομμάτι αυτού. Γι' αυτό και Τονίζεται το άρθρο 9, όλοι λένε να το χρησιμοποιήσουμε. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να σκεφτείτε πόσο πιέζεται έτσι το 9 και η οδηγία. Γιατί χρησιμοποιείται για κάτι που ειδικά για κάποια από τα πιλωτικά προγράμματα τώρα είναι σαφώς βιομηχανικές μεταφορές ανάπτυξης που χρησιμοποιούν πολύ ακριβή ηλιακή τεχνολογία. Ας το έχετε αυτό υπόψη σας και μην το παρακάνετε με το άρθρο 9. Τώρα τι σημαίνει το άρθρο 9. Υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ω κράτο μέλο σε μια χώρα εκτό Ένωση και το όφελο είναι ότι πρέπει να καταναλωθεί στην κοινότητα την οποία γίνεται. Και έχει μετά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτό το επιπλέον ε, κομμάτι ανασυνεώσιμη ενέργεια στο δικό σου ενεργειακό μείγμα. Έπειτα, Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειε το αν δίνεται άλλη βοήθεια στις συγκεκριμένε εγκαταστάσει. Το θέμα είναι τι καταναλώνεται. Τι καταναλώνεται σύμφωνα με την οδηγία. Υπάρχουν τρει απαιτήσει. Ένα αντίστοιχο ποσό ηλεκτρισμού έχει οριστεί στη συγκεκριμένη δυνατότητα διασύνθεσης από όλες τις υπεύθυνε ε, χώρες, δηλαδή χώρα προέλευσης, χώρα προορισμού και κάθε χώρα διέλευσης. Αν η χώρα που θέλει να ωφεληθεί από αυτή την πράσινο ηλεκτρισμό είναι πιο μακριά και υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη ενδιάμεσα. Αυτό το αντίστοιχο ποσό θα πρέπει να καταγραφεί στο σχέδιο ισορροπίας από την υπεύθυνη υπηρεσία στην ευρωπαϊκή πλευρά. Η συγκεκριμένη δυνατότητα και παραγωγή ηλεκτρισμού θα πρέπει να αναφέρεται στην ίδια χρονική περίοδο. Αυτή είναι η βάση. Αν επιτευχθούν αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, τέλεια. Όμως η πραγματική μεταφορά, και δεν έρχομαι σε κάποια θέματα που μπορώ μόνο να σας δώσω μια εικόνα, μια γεύση, Συνάδελφοι, όλοι μαζί συνεργαζόμαστε με στόχο να το πετύχουμε αυτό. Έχουμε δύο δικηγόρους, έχουμε τρεις απόψεις, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η πραγματική μεταφορά είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί πού θα καταγραφεί στο τέλος ε, της σύνδεσης. Η υποχρέωση καταγραφής θα πρέπει να διευκρινιστεί. Όμως η ίδια η διασύνδεση είναι ένα κομμάτι το οποίο υπόκειται σε διάφορες εθνικές νομοθεσίες και από τις δύο πλευρές της θάλασσας. Μπορεί δηλαδή να, θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο σύστημα επαλήθευσης και εδώ μπαίνει πολύ πολιτική, πολύ προπαγάνδα στη σημερινή συζήτηση που εγώ πολύ θα ήθελα να την ξεφορτωθώ γιατί χρειάζομαστε το χρόνο μας για άλλα πράγματα χρησιμότερα. Κάποιοι τώρα λένε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την προέλευση ως πιστοποιητικό. Η χώρα προέλευσης, όπως ξέρετε εσείς οι ευρωβουλευτές, είχαμε μια πολύ δύσκολη συζήτηση για τη χώρα προέλευσης με την Επιτροπή, γιατί η Επιτροπή Ήθελε να εκδώσει πράσινα επιστοποιητικά, μετά δέχτηκε ότι δεν ήταν αυτό, σωστό, μετά ακούσαμε για την εναρμόνιση, μετά μη εναρμόνιση κτλ. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την συμμόρφωση προς τους δασμούς. Είναι μόνο μια απόδειξη για το ότι πράσινη ενέργεια, πράσινος ηλεκτρισμός πάει από μια χώρα στην άλλη. Σύμφωνα με την οδηγία δεν μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρισμό που προέρχεται από τρίτη χώρα όμως. Οπότε κάτι που είναι δύσκολο και που κάποιοι λένε πως για προσχάριν της χρηματοδότησης να αφήσουμε την πράσινο ηλεκτρισμό που παράγεται μέσα στο μείγμα των ε, τρίτων χωρών να μπει μέσα στο πρόγραμμα και στο μείγμα του ε, κάθε κράτους μέλους. Ε, πρέπει να διαφοροποιήσουμε εδώ τι θέλει να κάνει το κράτος μέλος και τι μπορεί να κάνει η οδηγία. Και η οδηγία λέει πως αυτό δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη στόχων, διότι εκεί σαφώς λέει πως μόνο η ευελιξία στο άρθρο 9 ανάμεσα στο να επιτρέψει δηλαδή πρόσβαση σε ένα άλλο κράτος μέλος με οποιοδήποτε μηχανισμό, αυτό είναι που ισχύει. Και σαφώς δεν αναφέρει τρίτες χώρες. Η τρίτη χώρα δεν υπάρχει. Αυτό σημαίνει πως κάποιος ανταγωνιστής ή κάποιος άλλος μπορεί να πει όχι, δεν γίνεται άλλο να επεκτείνουμε την έννοια της οδηγίας. Γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να αποκαθιλωθεί, να απομυστικοποιηθεί ε, αν υπάρχει διμερή συμφωνία με μια τρίτη χώρα, με το Μαρόκο, για πρόσβαση στο σύστημα, ε, τίθεται βέβαια το ζήτημα του πώς θα και πάρουμε αυτό το όφελος. Μέσω στατιστικής μεταφοράς τελείως διαφορετικό σύστημα. Δηλαδή κάποια κάτι μέλη συνεργάζονται, ζητούν κάποιο αντίστοιχο πράσινη ενέργειας από κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να εισαχθεί. Ναι, ναι, το ξέρω πως ήδη έχω πολλά. Αλλά έχω κάτι ακόμα και θα τα αφήσω εκεί στην οθόνη. Υπάρχει ένας κατάλογος με τελίτσες για ερωτήματα σε σχέση με την ε, σύνδεση του πλέγματος, ε, Ποιε είναι οι διαδικασίε σύνδεση του πλέγματο στι τρίτε χώρε, αν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για την προώθηση και το σύστημα τη ε, νεώσιμη ενέργεια, ποια είναι τα τέλη, ποιο τα καταβάλει, πώ λειτουργεί αυτό το σύστημα, πώ γίνεται με το κράτημα των, εκπομπών, των, των μεταφορών κτλ. 40-50 ερωτήσει μόνο. Και όπω σα είπα είναι υπό εξέλιξη όλα αυτά. Δεν θέλω να φύγουμε από εδώ στεναχωρημένοι. Όχι. Γι' αυτό νομίζω συνδέεται με τα όσα είπε ο συνάδελφο από την Κομισιόν. Πρέπει να δουλέψουμε με διμερεί συμφωνίε, με την. Ανταλλαγή πληροφοριών. Το μπαλάκι είναι λοιπόν στο γήπεδο των κρατών μελών. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός η Ισπανία πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο για να γίνει αποδεκτή, για να βοηθήσει άμεσα τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε μπροστά και πρέπει να σκεφτούμε το 2020 να έχουμε ε, ε, μια ατζέντα πράσινης ενέργειας. Γιατί μετά το 2020 θα θέλουμε δεσμευτικού στόχους για το 2030. Και όπως είπαν και οι Ισπανοί συνάδελφοι από την RED, Εύκολο είναι να λέμε σταματήστε τον αέρα στην Ισπανία και θα το παίρνουμε από τη Βόρεια Αφρική γιατί είναι ένα-δυο λεπτά φθηνότερο. Δεν μπορούμε, μπορώ να πω και παραπάνω. Σταματήστε τη φωτοβολταϊκά στην Νότια Σουηδία ή στην ε, Γερμανία. Μα δεν ε, γι' αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε ένα σωρό συστήματα. Γι' αυτό η έκκλησή μου είναι να δουλέψουμε, δουλέψουμε σκληρά, αλλά να καταλάβετε ότι το άρθρο 9 είναι απλά ακόμα ένα εργαλείο. Ευχαριστούμε πολύ. Βρίσκομαι κάπως σε δύσκολη θέση, διότι συνήθως μόνο ε, οι ευρωβουλευτές μπορούν να θέσουν ερωτήσεις. Ε, είναι, λίγο, λοιπόν είναι λοιπόν λίγο περίεργο να δίνω το λόγο στον εαυτό μου. Ε, αυτό είναι λίγο το πρόβλημα των ακροάσεων που πραγματοποιούνται αργά την Πέμπτη το απόγευμα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να πάω στις διαπραγματεύσεις που σας είπα. Προτείνω λοιπόν πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του Κοινοβουλίου που ε, έκαναν δυνατή αυτήν την ε, ακρόαση. Ο πρόεδρος Ρόιλ εμπιστεύτηκε κάποιους ευρωβουλευτές ε, να εκπονήσουν το πρόγραμμα αυτό. Το προσωπικό μας, σας παρακαλώ σηκωθείτε να σας δούνε όλοι ποιος βρισκόταν πίσω από την οργάνωση της ακρόασης αυτής. Εγώ θα πρότεινα το εξής λοιπόν. έχουμε μια ομάδα ε, ε πολύ ανθρώπων με ε, εξαιρετικές ικανότητες και γνώσεις. Ε, ε, θα ήταν κρίμα να διαλυθεί πάλι η ομάδα. Θα πρότεινα κάποιος να πάει μαζί σας σε ένα μπαρ εδώ στην Πλάσου Λουξεμβούργκ. Σε μισή ώρα θα είμαι πάλι μαζί σας για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. θα παρακαλούσα κάποιον να, πάρει, να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό για μένα θα ήταν το